Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ξεκινάμε με το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Αν έχετε παρατηρήσεις ή προτάσεις, παρακαλώ να μου το πείτε. Αλλιώς θεωρούμε ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Τώρα, προτείνω να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα επιτρουσίας στην εμμυρίσια διάταξη, που είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου ΕΚΟΝ. Θέλω να σας ενημερώσω για το γεγονός ότι ο πρόεδρός μας σήμερα συμμετέχει στο τριμερή διάλογο σχετικά με τα μέτρα δημοσιονομικής ρύθμισης. Άπαξ και η συνεδρίαση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί του τριμερούς διαλόγου, θα έρθει και θα αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής μας εδώ. Θέλω όμως να σας διαβάσω αυτά που μου ζήτησε να σας ανακοινώσω εκ μέρους της. Έχουμε για σήμερα το απόγευμα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και όπως θα έχετε δει και από το δεικτικό χρονοδιάγραμμα που έχει κυκλοφορήσει, είναι απαραίτητο να τηρήσουμε το χρόνο για το κάθε σημείο. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μια ιδανική κατάσταση, αλλά επειδή έχουμε τεράστιο φόρτο εργασία, δεν έχουμε άλλη λύση. Γι' αυτό θα σας ήμουν ευγνώμων εφόσον όλοι σας, όλοι οι ομιλητές δηλαδή, στα διάφορα σημεία της ημερήσιας διάταξης, έχετε υπόψη στον περιορισμό αυτού του χρόνου. Δεύτερη ανακοίνωση. Σα έχω ήδη πει για την έκτακτη συνεδρίαση που προβλέπουμε για την 5η Ιουλίου της Επιτροπής μας, 7 με 9 ε, μετά το μεσημέρι. Ο Επίτροπος Όλη Ρεν στο μεταξύ μας επιβεβαίωσε ότι θα έρθει στην Επιτροπή μας το βράδυ και στην ίδια συνεδρίαση θα έχουμε και το σχέδιο για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μέσα στην Ευρωζώνη, που θα υποβληθεί από την εισηγητή μας, τον κύριο Φέο. Τρίτη ανακοίνωση. Ζητήσαμε άδεια για μια άλλη έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για την 5η 8 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί. Η μερίσια διάταξη θα συμπεριλάβει του οίκου αξιολόγηση κατά πάσα πιθανότητα και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το Solvency. Άλλες... Αυτές μάλλον ήταν οι ανακοινώσει που μου ζήτησε η Πρόεδρός μας να σας μεταφέρω. Τώρα, ερχόμαστε στον κύριο Αλγίδρα Σέμετα, που είναι επίτροπο για την Φορολογία και την Τελωνιακή Ένωση τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης. Θα μας παρουσιάσει τις κύριες προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, Θυμάμαι πόσο πολύ σας ε, ενδιαφέραν τα θέματα φορολογίας. Και γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα για να μοιραστώ μαζί σας τις φιλοδοξίες μου για τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πάνω σε μια κοινή, πιστεύω, μερίσια διάταξη. Επί τη αυτή, μάλιστα, θα σας υπογραμμίσω τα κύρια στοιχεία του νομοθετικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της φορολογίας. Η κρίση ανάγκασε τα κράτη-μέλη να ξαναδούν και να αναθεωρήσουν τις δικές τους οικονομικές πολιτικές. Η Ευρώπη θέλει ευημερία και έχει αντιληφθεί ότι χρειάζεται φορολογικές αλλαγές, ε, προσαρμογές σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν πόσο εξαρτώνται οι οικονομίες των κρατών μελών του ενός από το άλλο. Και είμαι πεπισμένος ότι ο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι αναγκαίο, ζωτική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαι έτοιμος να χρησιμοποιήσω ό,τι μέσα έχω στη διάθεσή μου για να διασφαλίσω όπου αυτό είναι αναγκαίο ότι οι εθνικές φορολογικές πολιτικές ε, συγκλίνουν. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο χώρο για να συζητήσει την ε, πολιτική της όσον αφορά τη φορολογία και γι' αυτό θα ήθελα τακτικά να έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας και να ανταλλάσσω απόψεις μαζί σας για αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι έχετε πολλά να προσφέρετε στη συζήτηση αυτή. Ελπίζω και σήμερα ότι θα έχουμε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στο και μου. Ενίσχυση του οικονομικού συντονισμού, για παράδειγμα, η συνεισφορά της φορολογικής πολιτικής στην ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας. Πρώτα απ' όλα, Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για το πόσο σημασία έχει η ποιότητα των εσόδων μας προκειμένου να πετύχει η στρατηγική μας εξόδο από την κρίση. Σήμερα που βρισκόμαστε σε τέτοιες δυσκολίες, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προκλήσεις προκειμένου να ετοιμάσουν τα προγράμματα τους φορολογικής πολιτικής. Κανείς ε, βέβαια δεν αμφισβητεί το θέμα της ποιότητας των δαπανών. Όμως, αν λάβουμε υπόψη μας ε, και το θέμα της, των εσόδων από τη φορολογία είναι και αυτό εξίσου σημαντικό, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ποιότητά του. Πώς λοιπόν θα αναθεωρήσουμε τα φορολογικά συστήματα, πώς θα τα διαμορφώσουμε έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε την απασχόληση και τις επενδύσεις και να έχουμε μια πιο πράσινη οικονομία που να βασίζεται στην κοινωνία της γνώσης. Όλα τα κράτη-μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν ποια θα είναι η δικιά τους προσέγγιση. Όμως είμαι πεπιδισμένος ότι 27 χώρες μονομερός και χωρίς συντονισμό, 27 διαφορετικές προσεγγίσεις σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε. Έχοντας αυτό υπόψη μας λοιπόν και ε, δουλεύοντας στην ανάλυση των φορολογικών προγραμμάτων και φορολογικών σχημάτων των χωρών μελών, θέλουμε να πετύχουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη καλύτερη φορολογική πολιτική και πρωτοβουλίε για το μέλλον. Για να πετύχουν οι συζητήσει αυτέ, έχω ήδη ξεκινήσει με μια ομάδα φορολογία τη οποία και προεδρεύω, και έχω ζητήσει από του Υπουργού Οικονομικών να ορίσουν έναν εκπρόσωπό του, έτσι ώστε να μπορέσουμε από κοινού να εξετάσουμε σε πολιτικό επίπεδο πώ μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο υπέρ μια ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική υπέρ τη ανάπτυξη. Και έτσι θα κοιτάξω και το θέμα του δημοσιονομικού τομέα προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε την έξοδο από την κρίση. Βέβαια, η πολιτική συζήτηση προχωράει με πολλά επίμαχα θέματα και πολλά παραμένουν σε κρεμότητα. Τα θεσμικά όργανα εξετάζουν κατά πόσε συναλλαγέ πρέπει να φορολογηθούν, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει από μόνη τη, πώ πρέπει να ε, κατανείμουμε στη συνέχεια τα έσοδα από έναν τέτοιο εκτακτοφόρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κάνει ένα πρώτο βήμα και ζήτησε να υπάρξει μια εισφορά τραπεζών που να μας ε, βοηθήσει να προχωρήσουμε κάτι το οποίο καλωσόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε το, ε, την, το ψήφισμα που πρότεινε η πρόεδρό σα τον προηγούμενο μήνα για να εξετάσουμε το θέμα της φορολόγησης των τραπεζών επίσης. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των ε, συζητήσεων θα καταλήξει κάπου στα μέσα της εβδομάδας και αυτό δείχνει τι τεράστιες προκλήσεις έχουμε μπροστά μας και ότι χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση. Τώρα μένει να δούμε κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να συνεχίσει μόνη της φορολογώντας ε, τον δημοσιονομικό τομέα. Αν θέλετε πρόοδο, πρέπει να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις που θα έχει ένας τέτοιος φόρος την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεύτερον, φορολόγηση για εφόρο ανάπτυξη. Είπαμε ότι θέλουμε να δώσουμε νέα όθηση στην ενία αγορά για να στηρίξουμε την αηφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της στρατηγικής μας για το 2020. Όπως υπογραμμίζει η έκθεση Μόντι πρόσφατα, χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία που θα βασίζεται σε μια εσωτερική αγορά η οποία θα λειτουργεί καλά και θα είναι ισχυρή. Καλές φορολογικές πολιτικές είναι βασικό θέμα για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας ώστε να συνεισφέρουν αυτές σε άλλους στόχους μας, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν πολλά εμπόδια στην εσωτερική αγορά ακόμα. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να βελτίσουμε την φορολόγηση έτσι ώστε να είναι πιο φθηνή η λειτουργία των επιχειρήσεων όταν αυτές δρούν διασυνοριακά. Θέλουμε επίσης να ασχοληθούμε και με τον πολίτη. Η έκθεσή σας της κυρίας Γκρέτς υπογραμμίζει ότι πρέπει στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς πρέπει να βάλουμε τους πολίτες που ζουν μέσα στην εσωτερική αγορά, την καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό και θέλουμε να άρουμε τα εμπόδια, τα φορολογικά, τα οποία δημιουργούν ε, συχνά προβλήματα για τους πολίτες μας. Να κοιτάξουμε τα δικά τους τα προβλήματα, διπλή φορολόγησης, διακρίσεων που γίνονται σε βάρος τους στη φορολογία. Αυτά είναι πράγματα που είναι από τις πρώτες προτεραιότητές μου. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Στις 27 Απριλίου ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση για να ρωτήσουμε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να μας μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την διπλή φορολογία κατά τις διασυνοριακές τους συναλλαγές. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή μια νέα δημόσια διαβούλευση που έχει να κάνει με διασυνοριακά ζητήματα όσον αφορά τον φόρο κληρονομιάς. Επίσης θέλουμε να εξετάσουμε την φύση και το εύρος των προβλημάτων αυτών. Και βάσει των αποτελεσμάτων θα προχωρήσουμε σε απαντήσεις. Όσον αφορά τώρα την ε, μείωση του κόστου συμμόρφωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέτυχε μια συμφωνία όσον αφορά τον ΦΠΑ. Και παρόλο που δεν πάει η συμφωνία αυτή όσο μακριά θα ήθελε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλα αυτά αποτελεί ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Για το μέλλον θα φροντίσουμε για δράσεις ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς στον τομέα της φορολογίας. Αυτό τι σημαίνει. Πρώτον, εναρμόνιση του εταιρικού φόρου, της βάσης εταιρικού φόρου. Θέλουμε κοινού ευρωπαϊκού κανόνες, ώστε έτσι να έχουμε λιγότερο κόστος, προκειμένου να ταιριάξουμε τα εθνικά συστήματα με άλλα συστήματα όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που δρούν σε περισσότερες από μία χωρε Δεύτερον, θα ξεκινήσω μία πράσινη βίβλο για την αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ με τον στόχο να έχουμε ένα πιο δίκαιο και ένα πιο καλό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και ένα πιο ισχυρό σύστημα για τα κράτη-μέλη. Τρίτον, Βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης θα προτείνω στο Σώμα των Επιτρέπων μία ανακοίνωση για να καθορίσουμε ένα πρόγραμμα δράσης καταπολέμησης των ζητημάτων που προκύπτουν από τη διπλή φορολογία και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με το φόρο κληρονομιάς, όπως επίσης κατάσταση ή άλλα ζητήματα ε, από τα οποία υποφέρουν οι πολίτες μας. Τέλος, πιστεύω πως ε, πρέπει να προχωρήσουμε στην πράσινη φορολόγηση για να συνδυαστεί αυτό με τους ευρύτερους ε, στόχους ε, της ε, κλιματικής αλλαγής και άρα θα αναθεωρηθεί και η φορολόγηση της ενέργειας. στο σώμα των επιτρόπων συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα με αυτό ακριβώς το αντικείμενο και φτάσαμε σε συνένεση στο ότι το τωρινό σύστημα δεν δουλεύει όσο καλά θα μπορούσε για να υποστηρίξει αυτούς τους κοινούς στόχους όπως η μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης και θα τα λάβω υπόψη όταν θα ολοκληρώσω τη μελέτη αντικτύπων που θα ολοκληρώσει αυτή την πρόταση την οποία σκοπεύω να καταθέσω στο μότρο δυνατόν. Τρίτον, η καλή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας. Θα ήθελα να τελειώσω, τε, τελειώσω λέγοντας πόσο σημαντικό να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να συλλέξουν τα έσοδά τους, ειδικά τώρα που η καιρή είναι δύσκολη. Προς αυτό το σκοπό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τον αγώνα της κατά της φοροδιαφυγής και να συνεχίσει να δίνει τον αγώνα καλής διακυβέρνησης διεθνώς. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το Συμβούλιο έφτασε σε μια συμφωνία για την σύσταση της Eurofisk, η οποία θα αποτελέσει έναν πολυμερή μηχανισμό καταπολέμησης της απάτης του ΦΠΑ. Σε διεθνές επίπεδο έχει σημειωθεί επίσης ε, πρόοδος με την ανακοίνωση για το φόρο και την ανάπτυξη που προωθεί τις αρχές ε, καλής διακυβέρνησης από τις όμονες χώρες. Επίσης, το τελευταίο κοφήν ζήτησε από την ε, Κομισιόν να ξεκινήσει συνομιλίες με την Ελβετία και το Λιχτενστάιν για να τις ενθαρρύνει να ε, εφαρμόσουν τον κώδικα καλή συμπεριφορά για το φορολογικό ανταγωνισμό. Ήδη ξεκινάμε συνομιλίε με την Ελβετία. Για το μέλλον είμαι πεπισμένο πως θα πρέπει να διατηρήσουμε τις προσπάθειές μας ε, κατά της ε, φοροδιαφυγής και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος για την καλή διακυβέρνηση στα φορολογικά το να επεκταθεί η αρχή του κώδικα συμπεριφοράς στις τρίτες χώρες δεν αρχεί. Το πεδίο εφαρμογή του ίδιου του κώδικα πρέπει να επανεξεταστεί σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Μία άλλη προτεραιότητα είναι να δούμε πρόοδο στις συνομιλίες με το ΕΚΟΦΗΝ για το λεγόμενο πακέτο καλής συμπεριφοράς που αφορά τη διοικητική συνεργασία και συμφωνίες καταπολέμησης απάτη με τρίτες χώρες. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσο αποτελέσματα όσο θα ήθελε και η ε, Προεδρία και η Κομισιόν. Η διαπραγματεύση είναι δύσκολος, όμως ε, θα συνεργαστώ με τη Βελγική Προεδρία για να συμφωνήσουμε σε αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, αναφέρθηκα στους τρεις πυλώνες ε, του φορολογικού μου προγράμματος και της πολιτικές μας για το 2010-2011. Υπάρχει νέα ορμή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής φορολογίας, δεδομένου του ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας εάν μείνουν τα πράγματα όσο έχουν ή αν δρούμε μόνοι μας. Εάν εκμεταλλευτούμε αυτή την ορμή, είμαι πεπισμένος πως μπορούμε να έχουμε ποιοτική φορολογία η οποία θα είναι δίκαιη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη. Οι δράσεις μου αυτό θα έχουν ως όραμα. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει και εσείς έχετε σημαντικό πολιτικό ρόλο να παίξετε με το να στηρίξετε εδώ στο Κοινοβούλιο και στις χώρες σας ε, το πακέτο αυτό ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτό το οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θεωρούν μια διάσταση ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να υπενθυμίσω συναδέλφους η, πως η Επιτροπή μας ε, διεξάγει δομημένο διάλογο με τους τέσσερις επιτρόπους τους κυρίους Σαλμούνια, Μπαρνιέ, Ρεν και τώρα τον κύριο Σέμετα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. to Mr. Κύριος Μπούλμαν έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτά τα οποία μας λέτε ακούγονται ωραία. Χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πιο σοβαρή συζήτηση για τη φορολογική πολιτική. Αυτό δεν αμφισβητείται. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εκτιμήσετε την κατάσταση μετά το, το ρόντο, το Σαββατοκυριακό που πέρασε και να τοποθετηθείτε εδώ στην Επιτροπή μας για το που βρισκόμαστε. Θα σας πω τι εκτιμώ εγώ. Δεν προχωρήσαμε σε κεντρικά ζητήματα της καταπολέμησης της κρίσης γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδείξαμε ενότητα και αποφασιστικότητα. Άλλοι που έχουν συμφέροντα τα δικά τους, όπως οι χώρες οι αναπτυσσόμενες, δεν βλέπουν γιατί να λύσουν τα δικά μας τα προβλήματα αν εμείς δεν είμαστε αρκετά ισχυροί. Και είπα δεν βλέπει γιατί πρέπει να λύσει μαζί μας ε, προβλήματα αν δεν υπάρχει ένα πακέτο όσον αφορά και το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης ε, του να δοθεί μια όθηση στην οικονομία. Οπότε απομένει σε εμάς να μην είμαστε αποφασισμένοι, να μην έχουμε κοινή θέση και αυτό ισχύει ειδικά για τα θέματα τα οποία ζήτησε από εσάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνετε μια πρόταση, είπαμε, ε, από την Επιτροπή μας, στην Ολομέλεια, με πλειοψηφία, πώς χρειαζόμαστε μία εκτίμηση του φόρου στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ως ένα στοιχείο πρόληψης της ε, κρίσης και ως μια βασική πηγή εσόδων των κρεωμένων προϋπολογισμών. Και ζητάμε από την Κομισιόν να κάνει μια ανάλυση και μια πρόταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε θα έρθει αυτή η πρόταση, πότε θα έρθει αυτή η ανάλυση. Είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο δεν φτάνουν πλέον οι δικαιολογίε. Βλάπτει αυτή η πολιτική την παγκόσμια οικονομία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε βήματα, πρέπει να λάβουμε δράση. Βασιζόμαστε, σα εκτιμούμε, αλλά πρέπει και εσείς να αντιδράσετε σε αυτά τα οποία δεν σας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απέτησε από εσά και αυτά ήδη εδώ και μερικού μήνε. Thank uh, Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και για τα σχόλιά σας. Uh, σε ό,τι αφορά τη σύνοδο των G20, πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε με θέληση και θέση για να συζητήσει ε, τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έγινε λοιπόν συζήτηση σε βάθος στην ομάδα των 20 με το εξής αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία παγκόσμια. On uh, financial sector. Για τη ε, φορολόγηση του χρωματοπιστωτικού λοιπόν, συστήματος υπάρχει διχογνωμία. Εμείς συζητούμε και θα προτείνουμε τη φορολόγηση των τραπεζών για μελλοντικά προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τώρα έχει έρθει όμως ο καιρός να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων ενδεχομένων προτάσεων φορολόγησης τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ενδυμάτων. Ήδη έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες μου να κάνω μια ακριβή εκτίμηση του φόρου του FTT ή άλλων φόρων χρηματικών συναλλαγών. FAT. Financial Activity Tax. Και αυτά τα συζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε σαφή αξιολόγηση. Ναι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα θέματα λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ενδιαφερμένους και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και να καταλήξουμε ε, σε οριστικά βήματα από εκεί και πέρα. Ε, και τώρα ο κύριος Λάμρεχτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Σεμετά και δεν το λέω προσωπικά, ξορίζω και πολλά από όσα είπατε, λέει ο κύριος Λάμπερτ στα αγγλικά. Πολλά από αυτά που μας είπατε μας χάιδεψαν τα αυτιά. Θα ήθελα ε, να πω ότι χαίρομαι που βλέπετε ότι έχει έρθει τώρα ο χρόνος να επιταχυνθεί η συζήτηση στην Ευρώπη για τα φορολογικά και συμφωνώ με την άποψη αυτή. Θα πρέπει να εντείνουμε και να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Και χαίρομαι επίσης και ε, για την προθυμία σας να συνεργαστούμε μαζί σας. Νομίζω ότι είναι ειλικρινής η προθέση σας. Το δείξατε από την πρώτη μέρα που ήρθατε στην ακρόαση όταν είχατε προταθεί για Επίτροπος και αυτό επίσης πολύ θετικό για μένα συμμεζόμαστε πολλούς από τους στόχους που παρουσιάσατε. Καλωσορίζουμε επίσης την ε, πρωτοβουλία που λάβατε για τη φορολογική πολιτική. Μου έκανε εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα που συζήτησα με τον Herman Van Rompuy και είδα ότι έχει και εκείνο μια ομάδα ε, κρούσης για τις δαπάνες ε, στα δημοσιονομικά που είναι τελείως απαγκιστρωμένη από αυτά που θέλετε εσείς να κάνετε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εσείς να σταματήσετε, όχι να συνεχίσετε την προσπάθειά σας, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι κάποια στιγμή οι δύο αυτές πρωτοβουλίες θα πρέπει να συναντηθούν, να διασταυρωθούν, διότι τι εστί προϋπολογισμός, έσοδα και δαπάνες. Και καλό είναι λοιπόν να ε, συνδυάσουμε αυτά τα δύο να συναντηθούν κάποια στιγμή. Λέει και ο κύριος ε, Ούρμαν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τη Σύνοδο των 20 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει μόνη της, θα πρέπει να ζητάει παγκόσμια λύση. Το ίδιο ισχύει και με την ε, ε, δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Το ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε παγκόσμια λύσει, αλλά γι' αυτό θα χρειαστούν χρόνια, για να μην πω ε, δεκαετίε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε μόνοι μα. Δεν θα πρέπει εμείς να αναλάβουμε ε, ηγετική θέση, να, ε, την πρωτοπορία και για το, τη φορολογία των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων και των συναλλαγών. Αυτό βοηθάει, δεν βλάπτει. Και τα ε, φορολογικά το ίδιο. Θα πρέπει και εκεί να είμαστε φιλόδοξοι. Τώρα, μιλήσατε για ζητήματα ανταγωνιστικότητας που συνδέονται με το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν προσπαθώ να το υποβαθμίσω, αλλά είδατε τι είπαμε για ε, το εμπόριο και την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Είπαμε ότι πάρα πολλέ επιχειρήσει αντιμετωπίζουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και χρειάζονται την προστασία μα. Αν όμω δείτε τα γεγονότα, είναι 5-6, δεν είναι και 162, ας πούμε, 100.000 επιχείρησεις. Να μην είμαστε υπερβολικά ε, προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Υπάρχει εσωτερική ζήτηση και αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και μας αρκεί αυτό για να επιβάλλουμε το φόρο. Τι θα γίνει τώρα με το εισόδημα ε, από τους φόρους. Πώς θα καταναμηθεί. Δεν έχουμε καταλήξει. Αλλά εάν επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος, θα πρέπει να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς ε, το προϊόν του φόρου αυτού και να δούμε τι θα ανακατανέμεται στα κράτη-μέλη, ίσως υπό τη μορφή της μειωμένης συνεισφοράς των κρατών των ιδίων προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ποιο τμήμα πηγαίνει ε, κατευθείαν στον προϋπολογισμό. Και έτσι θα έχουμε μία ε, κατάσταση που θα βγαίνουν κερδισμένοι και οι, οι δύο. Και τα κράτη θα έχουν περισσότερο κομμάτι από την πίτα και η Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον θα αυξηθεί το μέγεθός της. Το Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από δύο εβδομάδες ε, αυτούς τους στόχους της φιλοδοξίας και μπορεί ε, ο φόρος αυτός να βοηθήσει για την αναζωγόνηση και αναθέρμανση και την ανάκαμψη της οικονομίας. Μετά το καλοκαίρι λοιπόν θα συζητήσουμε, θα συνεισφέρουμε μαζί σας στην προσπάθεια αυτή και σας υποστηρίζουμε πλήρως. Ευχαριστώ. Ε, Thank you uh, Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και που καλωσορίζετε την δημιουργία αυτής της ομάδας φορολογικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει η πολιτική συζήτηση και η συζήτηση για τα φορολογικά εντό ένωση. Γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχουμε μια καλλιτεχνική συζήτηση, αλλά η πολιτική συζήτηση δεν, δεν προχωράει στα φορολογικά. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει μια σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδων. Γιατί δεν είναι μόνο έξοδα η φορολογική πολιτική, είναι και τα έσοδα. Έχει δύο πλευρές ο ισολογισμός και βεβαίως ε, πρέπει να υπάρξει μια, να γίνει μια μείωση των εξόδων αλλά με έναν έξυπνο τρόπο. Οπότε όσον αφορά το φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μετά τους G20 η κατάσταση έγινε σαφέστερη δηλαδή. Πρέπει να γίνει μια ανάλυση εις βάθος των πιθανών εναλλακτικών. Γιατί είτε μιλάμε για μετοχές και ομόλογα μόνο, είτε μιλάμε και για τα παράγωγα, γιατί τα έσοδα θα είναι πολύ διαφορετικά βεβαίως και θα εξαρτηθούν από τη φορολογητέα ύλη. Εγώ, εγώ είμαι ανοιχτό μυαλός άνθρωπος. Θα γίνει λοιπόν αυτή η ανάλυση, θα συζητήσουμε μαζί σας και με τα κράτη-μέλη και μάλλον σε τέτοια φόρα όπως την ομάδα οικονομικής πολιτικής με ποιο τρόπο πρέπει να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη αυτή δράση. Thank you. Mrs. Beres. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπέρες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν θα επαναλάβω όσα είπαν οι προλαλήσαντες που υπερθύμησαν πολύ καλά τι διακυβεύεται όσον αφορά τη φορολόγηση των ε, οικονομικών συναλλαγών. Πέρα όμως από την εντολή σας που είσαστε επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι έχετε και μια όλος ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτό το θέμα. Διότι αν δούμε την κρίση μέσα στην οποία έχουμε βουτήξει, Κυρία Μπερές, μπορείτε να σταματήσετε λίγο γιατί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τα αγγλικά. Δεν ακούγεται η αγγλική διερμηνία, λέει ο πρόεδρος διακόπτοντας την ομιλήτρια. Δεν ήξερα ότι είναι δύσκολο να μεταφράζονται τα γαλλικά στα αγγλικά, λέει η κυρία Μπερές. Αλλά όλο και κάτι καινούριο μαθαίνει κανείς. Για να ελέγξουμε, λέει ο πρόεδρος. Έχει βάλει το σωστό κανάλι. Α, τώρα είσαστε εντάξει. Εντάξει. Συγγνώμη κυρία Μπερές που σας διάκοψα, διευθετήθηκε το θέμα. Μπερές. Λοιπόν, λέω ότι δεν θέλω να επαναλάβω τόσο είπαν οι προλαλήσαντες για τα συγκεκριμένα θέματα εφαρμογής της μέτρου φορολόγησης των οικονομικών συλλογών, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σα, μια που είσαστε επίτροπος υπεύθυνο για πρωτοβουλίες σε αυτά τα θέματα, αλλά και μέλος του σώματος του Επιτρόπου. Γιατί βλέπετε σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη θέλουμε ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και πρέπει να υπάρχει πρωτοβουλία για το θέμα αυτό των οικονομικών συναλλαγών. Αναφερθήκατε στον πολίτη. Ε, λοιπόν, κύριε Επίτροπε, πάρτε μια πρωτοβουλία ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, Α μην είναι ευρύτερη από αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πρωτοβουλία. Να ξέρετε ότι έτσι θα βρεθείτε πιο κοντά στου Ευρωπαίου πολίτε και αυτοί θα σα καταλάβουν καλύτερα. Εξάλλου θα είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία για πολλούς και διάφορου λόγου που δεν είναι ανάγκη τώρα να επαναλάβω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να αντικαταστήσει αυτό το φόρο οικονομικών συναλλαγών. Είτε πρόκειται για τις οικονομικές συναλλαγές, για μας οι οικονομικές συναλλαγές έχουν, η φορολογισή τους δηλαδή, έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι ρυθμίζονται οι αγορές έτσι. Και δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έτσι μπορούμε να έχουμε έσοδα για να χρηματοδοτήσουμε πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε διακαώς. Συνεπώς, τα συμπεράσματα του G20 δεν μας καλύπτουν πλήρως. Σύντομα τα έχω κοιτάξει, αλλά δεν βλέπω πουθενά να αναφέρεται κάτι για τη φορολόγηση των οικονομικών συναλλαγών. Για το Ταμείο εδώ στο παράρτημα μόνο βλέπω, στο παράρτημα 1, έτσι ασαφώς κάτι να αναφέρεται στην παράγραφο 21, που δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο όμως σε σχέση με τις προσδοκίες μας. Και έπειτα στα συμπεράσματα της ομάδας των 20 υπάρχει ένα θέμα το οποίο φαίνεται είναι της μόδας, μάλλον ήταν της μόδας, δεν είναι πια, ενώ για προηγούμενες συνεδριάσεις του G20 ήταν θέμα και είναι η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Δεν είναι όμως πια φαίνεται καθόλου της μόδας σε τέτοιο βαθμό που το G20 δεν το αναφέρει καν. Ακόμα μάλιστα και όταν ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης γιατί ξέρουμε τι ρόλο παίζουν οι φορολογικοί παράδεισοι που εμποδίζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν έσοδα πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξή τους. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω και τρία άλλα πράγματα εφόσον μου επιτρέπει ο Πρόεδρος. Πρώτον, σας άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση να αναφέρεστε στην ιδέα του φόρου για τις επιχειρήσεις. Στην αρχή της εντολής σας δεν αναφερθήκατε σε αυτό. Είναι ένα δύσκολο θέμα, σκληρό, αλλά ζωτική σημασίας. Ακόμα και με το πακέτο Μόντι. Αλλά θέλω πιο συγκεκριμένα να μου πείτε σε τι βάση θα κάνετε αυτή τη δουλειά θα χρησιμοποιήσετε εργασίες που έχουν γίνει από τον προκάτοχό σας. Για δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες επί της ουσίας για αυτό το θέμα και πείτε μας σε τι βαθμό, κατά τη γνώμη σας, η υπόθεση αυτή πρέπει να συνδεθεί με άλλες πτυχές του πακέτου Μόντι. Γιατί εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική. Το πακέτο Μόντι έχει διάφορα πολύ φιλελεύθερα στοιχεία που θα προχωρήσουν ε, με φοβερή ταχύτητα, τρένο υψηλή ταχύτητας και υπάρχουν άλλα στοιχεία σχετικά με τη φορολογία που θα πάρουν τον καρβουνιάρη. Θα πηγαίνουν πάρα πολύ σιγά και δεν θα προχωρήσουν με τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Δεύτερο ερώτημα. Μπορεί να μην σας άκουσα πολύ καλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν αναφερθήκατε στα φορολογικά συστήματα που έχουν να κάνουν με ε, πληρωμές σε μικρά χρονικά διαστήματα. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό. Τέλος, στην ομάδα εργασίας υπό την προεδρία του κυρίου Φαν πολλά αναφέρονται για κυρώσεις που θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη, τα οποία παρεκκλίνουν από τους κανόνες που έχουν αποφασιστεί. εδώ και λίγο καιρό με διάφορους παρατηρητές προτείνουμε να σκεφτούμε ευφυείς κυρώσεις. Αντί δηλαδή να χτυπήσουμε τον άταχτο, να βρούμε άλλους τρόπους για να το συμμορφώσουμε. Για παράδειγμα, μια χώρα η οποία έχει υπερβολικό έλλειμμα και που δεν τηρεί τους κανόνες, να αυξήσει το ΦΠΑ, ε, να έχει ένα φόρο για το διοξείδιο του άνθρακα, περιβαλλοντικό φόρο. Από ό,τι έχω καταλάβει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται τέτοιες ιδέες. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτές τις ευφυείς κυρώσεις και αν τα έχετε συζητήσει καθόλου με τον Επίτροπο Λιρέν. Απάντηση ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Mm. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. για τις οικονομικές συναλλαγές και την φορολόγησή τους ή και τις δραστηριότητες, συναλλαγές έχουν τα υπέρ και τα κατά τέτοιου είδου μέτρα. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε πολύ προσεκτικά τις διάφορες περιπτώσεις, ποιες συναλλαγές δηλαδή θα φορολογούμε και στη συνέχεια να το συζητήσουμε αυτό και με εσά και με όλους τους εμπλεκόμενους για να βρούμε πώς είναι καλύτερα να προχωρήσουμε. Πάντως, από αυτού, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα των ε, αμοιβών, η δικιά μας η ανάλυση και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνουν ότι καλύτερα θα ήταν να έχουμε φόρο, φόρο ε, δραστηριοτήτων, οικονομικών δραστηριοτήτων, γιατί έτσι με το σύστημα αυτό έχουμε καλύτερη απόδοση και μπορούμε καλύτερα να σχεδιάσουμε αυτό το φόρο εφόσον ε, δεν υπάρχει αρκετό ρευστό, μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Για το CCTB. Εδώ γίνεται αξιολόγηση επιπτώσεων και αυτό ξέρετε επειδή ζήτησα από τις υπηρεσίες να κοιτάξουν λίγο την πρόταση αυτή όχι μόνο από την πλευρά των πολυεθνικών, αλλά και από την πλευρά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε να απλοποιήσουμε την πρόταση με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε διεθνές επίπεδο. Αυτή την εποχή ετοιμάζουμε την αξιολόγηση επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη κάποια ζωτικά μεγάλα θέματα. Να υπάρχει κοινό, κοινή βάση τελικού φόρου, παγιωμένη και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, μια τέτοια βάση θα είναι σε θελοντική βάση ή πρέπει να είναι υποχρεωτική. Αυτές οι αξιολογήσεις γίνονται λοιπόν αυτή την εποχή. Πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά αυτή. Οπότε τον επόμενο χρόνο θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Την επόμενη χρονιά λοιπόν. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011. Για το θέμα τώρα των κυρώσεων, την Τετάρτη το Σώμα των Επιτρόπων θα συζητήσει πρόταση της Επιτροπής για την χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Όλυ Ρεν, πρέπει να σας πω. Το δικό μου το χαρτοφυλάκιο είναι συμπληρωματικό με το χαρτοφυλάκιο του Όλυ Ρεν που ασχολείται με την οικονομική διακυβέρνηση και έχετε δίκιο ότι ένα σύστημα κυρώσεων πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η παρέμβαση να γίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να μην περιμένουμε να φτάσουμε σε καταστάσεις όπου τα κράτη μελίδη βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε μεγάλες δυσκολίες. Ο Όλη Ρεν ετοιμάζει μια σχετική πρόταση. Thank Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Κλούτε. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, και εγώ ήθελα να σα ρωτήσω κάτι για τον φόρο των συναλλαγών. Έγιναν πολλές ερωτήσεις. Ε, μας είπατε αρκετά πράγματα, οπότε δεν θέλω να επαναλάβω την ερώτηση. Απλά συμφωνώ με τους προλαλήσαντες με το ενδιαφέρον που επέδειξαν και αυτό δείχνει πως ε, το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για αυτό το φόρο και για το τι θα γίνει. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω πως ε, εμείς ε, η ομάδα μου το υποστηρίζει και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κάτι σε αυτό το τομέα, αυτό θεωρούμε εμείς. Ήθελα να το πω αυτό σήμερα. Είχαμε γρήγορη αντίδραση όσον αφορά την Ελλάδα, όσον αφορά άλλε χώρε, όταν μιλάμε για την εξυγίανση του προπολογισμού και το ξεκαθαρίζουν αυτό νομίζω οι πολίτες πώς θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτοί. Οι δε τράπεζες όχι. Και όπως είπε και η Περβάνς, εάν είναι να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά την κακή οικονομική κατάσταση δεν μας μένει και πάρα πολύ ε, χρόνος. Πρέπει να συνεισφέρουν και ουσιαστικά οι τράπεζες στη χρηματοδότηση της κρίσης. Το ένα είναι αυτό που ήθελα να τονίσω και να πω. Το δεύτερο είναι πως τις τελευταίες μέρες στις γερμανικές ημερίδες διαβάσαμε πως στη Ρουμανία θα αυξηθεί κατά 5% ΦΠΑ. Πώς το εκτιμάτε αυτό. Αυτό κατά την άποψή μου σημαίνει πως ακριβώς οι άνθρωποι που έχουν χαμηλό εισόδημα πλήττονται δυσανάλογα για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και όχι οι τράπεζες που προκάλεσαν αυτή την κατάσταση. Να τονίσουμε αυτό. Και οικονομικά νομίζω είναι προβληματικό αυτό, αυτή η αύξηση του ΦΠΑ γιατί βεβαίως ε, δεν εξελίσσεται έτσι και η εσωτερική αγορά. Γιατί είπαν και οι προλαλήσαντες πως πρέπει να έρθουν και η κυρία Περβάνος πως πρέπει να έρθουν οι πολίτες και κοντά στην Ευρώπη. Δεν νομίζω να γίνει αυτό με την αύξηση του ΦΠΑ. Είναι ιδιαίτερο προβληματικό. Θέλω τώρα, με περιπτώσει, να ακούσω τη δική σας την άποψη. Ε, ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Ανέφερα ήδη αρκετές φορές πως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση το συντομότερο δυνατόν για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις ε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για το ΦΠΑ. Ξέρετε πως στο επίπεδο της Ένωσης έχουμε κάποια ελάχιστα, το ελάχιστο είναι 15% και δεν υπάρχει μέγιστο ποσοστό ΦΠΑ, αν και υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, πως το μέγιστο θα πρέπει να είναι ένα 25%. Οπότε εντό αυτού του πλαισίου τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να ρυθμίσουν το επίπεδο της φορολογίας. Και δεν είναι μόνο η Ρουμανία. Και άλλες χώρες νομίζω αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες ε, στην ε, δημοσιονομική τους ε, πολιτική. Προτείνουν λοιπόν να ανέβει το επίπεδο του ΦΠΑ. Ε, η χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα ανέβασε το ΦΠΑ από το 18% στο 21%. Οι δε γειτονικέ χώρες ακόμη ψηλότερα. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πως η φορολογητέα ύλη του ΦΠΑ είναι ευρύτατη, η φορολογική βάση και μία αύξηση του ΦΠΑ κατά 1% δημιουργεί πολύ σημαντικά έσοδα για τα κράτη-μέλη. Ε, Βεβαίω αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε για την ε, αντίστροφη αναλογικότητα του φόρου, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα και τα κοινωνικά ζητήματα μέσω των κοινωνικών πολιτικών τους. Πολιτικών που εφαρμόζουν. Αλλά ναι, είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους... Νομίζω πως η ομάδα φορολογικής πολιτικής είναι το βήμα εκείνο στο οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε τις πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά το φορολογικό τομέα και να ανταλλάξουμε και βέλτιστες πρακτικές και χείριστες πρακτικές για να διδαχτούμε και από τα καλά και από το όχι, τα όχι τόσο καλά. Από αυτά τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη. Και επειδή η πλειοψηφία των κρατών μελών χρειάζεται περισσότερα φορολογικά έσοδα, η συζήτηση αυτή και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα είναι χρήσιμη για να σχεδιάσουμε και μια έξυπνη στρατηγική εξόδου και για τα έξοδα και για τα έσοδα. Okay. Thank you. Now the... Ευχαριστώ. Η κυρία Ισαΐα τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζουμε η φορολογική πολιτική είναι από τα ουσιαστικότερα εργαλεία και από τους ε, τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας να υλοποιούμε τις ε, οικονομικές πολιτικές στα διάφορα κράτη-μέλη. Και να ξεπερνούν τα κράτη τα ελλείμματα του προπολογισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε ως βασικό πόρο το φόρο προστιθέμενης αξίας. Σε περίοδο όμως κρίσεων αυξάνεται ε, η πίεση να αποκτήσουμε ενιαία και κοινή οικονομική πολιτική. Εσείς το συζητάτε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω υπόψη μου εδώ το Φιλανδό Επίτροπο τον Όλι Ρεν και σας ρωτώ, μακροπρόθεσμα έχετε κανένα σχεδιασμό για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε συγκρούσεις εθνικής κυριαρχίας. Δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια ανησυχούν με τις εξελίξεις αυτές που βλέπουν στην οικονομική πολιτική και στη φορολογική όμως. Και θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το επίπεδο κοινή φορολόγησης. Ξέρω ότι ήδη κάποιες χώρες προβληματίζονται και κοιτούν ποιους φόρους μπορούν να αυξήσουν. Τις περισσότερες φορές είναι ο ΦΠΑ βέβαια. Είναι όμως πολύ χαμηλή η συλλογή των φόρων, γιατί μεγάλη η φοροδιαφυγή. Σε ορισμένα μέρη είναι μέχρι και εθνικό άθλημα. Έτσι λοιπόν Καλή αύξηση των φόρων, αλλά με τους έμεσους φόρους δεν καλυπτόμαστε και όλο και περισσότερο αυξάνεται η φορολόγηση της εργασίας ε, ε, γιατί είναι πιο εύκολο να συλλέγονται οι φόροι. Από εκεί και είναι μεγαλύτερη η φορολογική βάση. Πώς μπορούμε στο μέλλον λοιπόν να βελτιώσουμε τη δράση μας και την ποιότητα των φορολογικών μας συστημάτων. Πώς το βλέπει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθήσαμε, Φερρυπίν, να συνεργαστούμε για να ξεπεράσουμε για να... τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Πώς γίνεται όμως αυτό, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα καλύτερα τη συνεργασία αυτή και να εξηγήσουμε το φορολογικό στους πολίτες. Σε πολλά κράτη είπαμε ότι αυξήθηκε πρόσφατα ο ΦΠΑ. Οι συντελεστές δηλαδή. Ο τομέας όμως των υπηρεσιών και τομείς με ένταση εργασία τελικά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Γιατί υπάρχει και άλλο κόστος το οποίο δεν έχει συνυπολογιστεί. Δεν αρκεί να αυξηθεί η ΦΠΑ. Έρχεται να προσθεθεί μετά το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών. Ε, πράγμα που πιέζει, πολύ συμπιέζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσει Uh, uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Για την ενισχυμένη οικονομική συνεργασία και διακυβέρνηση. Κρίσιμο, πολύ κομβικό αυτό που λέτε. Και θα έπρεπε πραγματικά να ζητήσουμε την κατάλληλη ισορροπία, χωρίς να υπονομεύουμε την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών, να διατηρούν την αυτονομία τους στη χάραξη πολιτικής δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε βέβαιοι ότι οι πολιτικές αυτές είναι βιώσιμες. Από πλευράς, αν θέλετε, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και μακροοικονομικής σταθερότητας. Εν γέννη. Για τη φορολογία γνωρίζετε ότι στην Ευρώπη στους έμεσους φόρους έχουμε ένα σύστημα. Βέβαια πάντα χωρούν βελτιώσεις ε, τα πράγματα και υπάρχει και ανάγκη βελτιώσεων ε, άλλωστε στην άμεση πλέον φορολογία. Τι σας προτείνω λοιπόν. Εναρμόνιση ε, του φόρου των επιχειρήσεων, διότι αυτό έχει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της εσωτερικής ενιαίας αγοράς. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πέραν αυτού για να εναρμονίσουμε συντελεστές φορολογικούς σε χωράφια κυριαρχία των κρατών μελών, στους άμεσους φόρους, επαναλαμβάνω. Το βασικό εδώ ζήτημα δεν είναι η εναρμόνιση, αλλά ο καλύτερος συντονισμός. Τι θέλει ο καθένας να εφαρμόσει ο σύστημα, τα κράτη-μέλη με την ομάδα αφορολογικής πολιτικής να συντονίζονται και να διδάσκονται το ένα από το άλλο. Να είναι τα συστήματα πιο ευφυή και ε, προσανατολισμένα προς την ανάπτυξη για τη συλλογή τώρα των φόρων και τη φοροδιαφυγή είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεων. Και ελπίζω να ληφθεί η απόφαση και να βοηθήσει η απόφαση ε, ίδρυσης του οργανισμού Eurofisk για το ΦΠΑ. Βεβαίω ξέρετε ότι όλα αυτά χρειάζονται κάποιο χρόνο για να στηθούν και να αρχίσουν να λειτουργούν. Για πιο γρήγορη ανταλλαγή ε, πληροφόρηση των κρατών μελών. Διασυνοριακή συνεργασία. Συνεργαζόμαστε και με την Όλαφ, ας πούμε, για τα ζητήματα λαθρεμπορίου ε, γάρων και άλλων ειδών που υπόκειται σε ε, ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και η συνοριακή έλεγχη είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και πολύ σύντομα θα εξαγγείλουμε ορισμένες δράσεις στον τομέα αυτό. Ε, για το θέμα λοιπόν του ΦΠΑ και τους συντελεστές ε, φορολόγησης και το επίπεδο φορολόγησης σε τομείς ε, με ένταση εργασίας. Γνωρίζετε ότι η αντίστοιχη οδηγία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να υιοθετούν μειωμένους συντελεστές για τομείς ε, υπηρεσιών με ένταση εργασίας. Εναπόκειται όμως στα κράτη-μέλη προφανώς να το πράξουν, όχι σε εμά. Αν ζητάτε την προσωπική μου άποψη, για το ΦΠΑ και τις εξαιρέσεις ή τους μειωμένους συντελεστές. Δεν είμαι ένθερμος υποστηρικτής αυτών των μέτρων. Νομίζω ότι ο ΦΠΑ είναι πολύ καλός φόρος ε, για το σκοπό που δημιουργήθηκε. Βεβαίως τα κράτη-μέλη έχουν ε, το δικαίωμα, όπως σας είπα, και την επιλογή μέσα στο πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας να εφαρμόσουν μειωμένους συνταλιστές. Και στα παραρτήματα θα το βρείτε αυτό της οδηγίας. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπασέσκου. Thank you so much. Uh, Commissioner... Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον τελικό καταναλωτή των τραπεζών, δηλαδή από ό,τι κόστος επιβάλλεται στις τράπεζες, πώς θα φροντίσουμε να μην το αναλάβει τελικά ο καταναλωτής στις πλάτες του αυτό το βάρος. Θέλω, ειδικά για τη Ρουμανία, που αναφέρθηκε ο συνάδελφος, να του πω ότι εμείς αυξήσαμε το ΦΠΑ σύμφωνα με τη συμφωνία που είχαμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή ήταν μία, ε, ένα από τα πράγματα που ζήτησαν και συμφωνήσαμε μαζί τους. Την πήραμε λοιπόν την απόφαση αύξησης του ΦΠΑ, διότι πρώτα απ' όλα τα μέτρα ήταν να μειωθούν κατά 15% οι συντάξεις και οι μισθοί 25% Κάτι που απορρίφθηκε όμως τελικά από το δικαστήριο. Οπότε η τελική λύση ήταν η αύξηση του ΦΠΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ναι, ήταν ε, σχόλιο πιο πολύ το δεύτερο. Λοιπόν, το θέμα που θέσατε για την ε, μεταφορά του φόρου και του κόστου του, αν τελικά δηλαδή θα το αναλάβει στις πλάτες του καταναλωτής. Όντω αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε, να το εξετάσουμε, αναλύοντα τις επιπτώσεις, τον αντίκτυπο επιπτώσεων που θα έχει μια τέτοια φορολόγηση, ένα τέτοιο φόρος στι τράπεζε. Όντω πρέπει να δούμε τι επιπτώσει θα είχε ένα τέτοιο μέτρο πάνω στου καταναλωτέ. αν προχωρήσει μια τέτοια πρόταση, πρέπει να το δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη στην ε, μελέτη αντικτύπου. Αν το θέμα της ρευστότητας στην αγορά αντιμετωπίζεται έτσι. Είναι και αυτό ένα δύσκολο θέμα και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις δεν είναι εύκολο να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που σχεδιάζουμε τις προτάσεις μας. Διότι δεν μπορούμε με ένα μέτρο να αντιμετωπίσουμε όλες τις αρνητικές πτυχές. Κάθε πρόταση μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες και αργότερα θα φανεί αυτό, ότι έχουμε κάνει λάθος δηλαδή. Γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί, δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη με τις προτάσεις μας. Όταν πρόκειται για κάτι τόσο πολύ σημαντικό όπως είναι αυτό, ο φόρος δηλαδή για τις οικονομικές δραστηριότητες ή τις οικονομικές ε, συναλλαγές, θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για το ΦΠΑ άκουσα τα σχόλιά σας και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το ποσοστό ΦΠΑ είναι ένα θέμα που αποφασίζει το κάθε κράτος μέλος. Άρα η Ρουμανία στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνει την απόφασή της βάσει της οδηγίας βέβαια, αλλά για τα ποσοστά αποφασίζει η Ρουμανία. Αν ένα κράτος μέλος θέλει πάνω από 15%, 20% είναι απόφαση του κράτους μέλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Άλλες ερωτήσεις παρακαλώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τότε επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω συνάδελφοι, αλλά και σε εσά κύριε Επίτροπε, ότι σε συνάντηση των συντονιστών της Επιτροπής μας, της ΕΚΟΝ, αποφασίσαμε για τις εξής προτεραιότητες στον τομέα 2010-2011. Το πρώτο είναι αξιολόγηση επιπτώσεων όσον αφορά τον φόρο στις οικονομικές συναλλαγές, κάτι το οποίο το συζητήσαμε και εδώ μαζί σας. Αναθεώρηση επίσης του ενεργειακού φόρου, της οδηγίας για τον ενεργειακό φόρο. Ανακοίνωση για την φορολογία και την ανάπτυξη, ένα ελάχιστο, έχει ήδη γίνει. Πρόταση για το ΦΠΑ στα vouchers, πράσινη δήλωση για μια νέα στρατηγική ΦΠΑ, ανακοίνωση για μια φορολογική πολιτική πρώτο πολίτης, νομοθετική πρόταση επίσης για μια παγιωμένη βάση εταιρικού φόρου και εδώ θέλω να σας ρωτήσω κύριε πίτρο, πώς θα μπορούσατε να μας δώσετε λεπτομέρειες για αυτό το σημείο, για την βάση αυτή την κοινή εταιρικού φόρου. Στη συνέχεια, Έχουμε άλλες προτεραιότητες για την ανακοίνωση όσον αφορά τη μελλοντική στρατηγική ΦΠΑ για το 2011. Ανακοίνωση επίσης για τον συντονισμό των ε, φόρων κληρονομιάς και αναθεώρηση της οδηγίας για πληρωμές που γίνονται μεταξύ εταιριών διαφορετικών χωρών ε, μελών. Αν θέλετε μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες για, αυτό, για αυτή την βάση εταιρικού φόρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πως ε, ο προβληματισμός ε, και το πρόγραμμα της Επιτροπής συμφωνεί με το πρόγραμμα της Κομισιόν στον τομέα της φορολογίας και ελπίζω έτσι να έχουμε καλή συνεργασία. η την κοινή αυτή φορολογική βάση πρέπει να γίνει η τελική μας αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του έτους. Ανάλογα λοιπόν με το τι θα προκύψει από την αξιολόγηση αντικτύπου θα κάνουμε μια πρόταση αρχές του 2011. Και όπως σας είπα υπάρχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις. όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου και αφορούν είτε την κοινή φορολογική βάση είτε την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση και αν πρόκειται για ενοποιημένη φορολογική βάση ε, αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Αυτές είναι οι εναλλακτικέ λύσει οι οποίες εξετάζονται αυτή τη στιγμή από τις υπηρεσίε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είμαστε ιδιαίτερα που ήρθατε εδώ πέρα και θα σας προσκαλέσουμε βεβαίως και κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, ε, δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε μέχρι, μέχρι τις 4 και 30 γιατί ε, δεν έχουμε συγητές και εισηγητές, δεν είναι εδώ κανείς για τις εκθέσεις ε, που πρέπει να συζητήσουμε. Οπότε θα επαναληφθεί η συνεδρίαση στις 16.30. Ευχαριστώ. Right. We are resuming the meeting. Λαμβάνεται συνεδρίαση. And we are at point four. Είμαστε στο σημείο 4. Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Um, ο κύριος ε, Καράς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο πριν την ψηφοφορία. Ουσιαστικά, στη συζήτηση στην Ολομέλεια, μας ε, απασχόλησαν και θέσαμε και τις προϋποθέσεις για τη Eurostat, μια προφορική ερώτηση και με ένα ψήφισμα στη συνέχεια που εγκρίναμε στην Ολομέλεια στις τροπολογίες και στην αξιολόγησή τους. Εμπνεύστηκα από το ψήφισμα και μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που λειτουργήσαν αυτή τη φορά οι άτυποι διαβλή και το Συμβούλιο αποδυνάμωσε λιγότερο την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής από όσο είχαμε λόγους να φοβούμαστε. Η πρώτη άμεση αντίδραση για την Ελλάδα ήταν η αφορμή, γιατί είχαμε επί σειρά ετών ε, πλασματικά στοιχεία που είχαν σφρίση χωρίς αντίδραση της Eurostat και στο μέλλον δεν θα πρέπει να επιτρέπονται τέτοια φαινόμενα. Ε, ε, θέλω να μακρηγορήσω. Γνωρίζετε τι προτείνουμε και έχουν κατατεθεί τροπολογίες και σήμερα. κατά την άποψή μου, δέχομαι όλες τις επιθυμίες τροποποίηση με δύο εξαιρέσεις. Έχω παντού θετικό πρόσημο, εκτός από δύο, όπως σας είπα, γιατί κατά την άποψή μου αυτές οι δύο είναι προβληματικές. Η μία είναι 23 και η τελογική σκέψη του συναδέλφου Πόγκρος με μεγαλύτερη συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά την απόψή μου και μετά από συνεννόηση με τη Eurostat, αυτά είναι η νομοθεσία και δεν υφίσταται κανένας λόγος ε, των υστέρων να τα προσθέσουμε. Και θα πρότεινα στην τροπολογία λοιπόν Άριος Πόγκρος να καταψηφίσουμε για την αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη που να σας πω ποια είναι, είναι παριθμό 14. Επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά έχει λυθεί αυτό το θέμα νομικά. Μας τα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα. Στη συνέχεια έχουμε το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το αίτημα δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία στην Ολομέλεια κατά τη ψήφιση του ψηφίσματος. Γι' αυτό ε, το συζήτησα με το συντάκτη της νομοδότησης και την ομάδα των φιλελευθέρων που επιθυμούν και οι δύο και το λέω ειλικρινά να γίνει εξεταστική επιτροπή στο κοινοβούλιο. Και κανόνισα με τον συντάκτη μια προφορική τροπολογία που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει και τα λοιπά τα στατιστικά στοιχεία και να σβήσουμε το responsible parties για να μπορέσουμε να ε, συμφωνήσουμε όλοι με την τροπολογία αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ζητάμε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας ενημερώσει ξεκάθαρα να ερευνήσει και να καταλήξει θετικά ε, σε ποια λάθη έγιναν στο παρελθόν, παραλήψεις, ε, ολιγορίες και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χρειάζεται εξεταστική επιτροπή στο Κοινοβούλιο. Τώρα ε, είναι η σειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σας προτείνω λοιπόν να διαγράψουμε αυτές τις τέσσερις λέξεις για να μπορέσει να ψηφίσει η ε, Επιτροπή μας, οπότε και θα καταπέσει η τροπολογία υπαριθμών 9. Και όλες τις άλλες μπορούμε να τις ψηφίσουμε θετικά, να τις υπερψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Και για την προθυμία σας που δεν επιζητήσετε τη σύγκρουση αλλά τη συνένεση για να λύσουμε το ε, θέμα αυτό και να ενισχυθεί το Κοινοβούλιο και σε σχέση με τη Eurostat. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρας. Θέλει κανείς και ο να λάβει το λόγο. επειδή είμαι και εγώ σκιώδης εισηγητής, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, γιατί από πολύ νωρί άρχισε διαπραγματεύσει με τους σκιώδης εισηγητές που καρποφόρησαν διαπραγματεύσεις αυτές. Όπως βλέπετε συμπίπτουμε πάρα πολύ. Η πλειοψηφία των ε, τροπολογιών μας βρίσκει σύμφωνος. Σε σχέση με αυτό το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Κάρας, βεβαίως είμαστε όλοι υπέρ της διερεύνησης της καταστάσεως και ας βρουν ό,τι βρουν. Ε. Δεν θα πρέπει από τόσο νωρίς να στιγματίζουμε κάποιον και να προωθούμε φόβους και ανησυχίες. Ας τώρα αφήσουμε ε, το θέμα αυτό στη Eurostat να το εξτάσει, να το διερευνήσει, να κοιτάξει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, γιατί προσφέρεται ως μέσο διερεύνησης και μετά είδομεν. και στη συνέχεια αργότερα θα ψηφίσουμε και ελπίζω να υπερψηφιστούν οι τροπολογίες. Καλώς. We now come to... Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 5, η χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η εισηγητής είναι ο Τόμας Χέντελ. Ε, Κύριο Κλούτε θέλει να πει κάτι. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος του Τόμας Χέντελ, ο οποίος είναι άρρωστος αυτή την εβδομάδα. Δεν μπόρεσε να έρθει, μου ζήτησε να πω κάποια λόγια, εάν μου το επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστεί για την καλή συνεργασία. Υπήρχαν μια σειρά τροπολογιών που δεν συνέκλυναν όλες. Μετά έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε πέντε συμβαστικές λύσεις που δέχεται και η πλευρά μας και ελπίζουμε να βρουν κάποια πλειοψηφία ήδη από αυτό το γύρο. Δύο σημαντικά ζητήματα υπάρχουν από πλευρά μας. Συμβαστικέ βεβαίω προτάσει προτάσεις οδήγησαν στο ότι κάπως εξασθένησαν οι προτάσει του εισηγητή, αλλά βεβαίω αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτές τις περιπτώσεις και όλοι κάτι συνεισέφεραν. Ουσιαστικό είναι αφενός ε, αυτό το οποίο είναι η συμβαστική λύση Β, όπου λέγεται πως ζητάμε από την Κομισιόν να σκεφτεί τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις ε, που μεταφέρουν ε, τις ε, δραστηριότητες στο εξωτερικό και πώς θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση γιατί βεβαίως αυτές προκαλούν και την ανεργία και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό πως θα πρέπει να γίνει αυτό ένα μέσο αναδιάρθρωσης, όχι μόνο ένα μέσο στήριξης, αλλά να πιέσουμε ε, έτσι ώστε η Κομισιόν να καταθέσει κάποιες προτάσεις για το πώς θα έχουμε μια διαρκή, διαρκή αναδιάρθρωση της οικονομίας και αηφόρο. Και ένα τρίτο σημαντικό θέμα το οποίο οπωσδήποτε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα συνδικάτα είναι το αίτημα προς την Κομισιόν να σκεφτούμε πώς ε, μπορούν να απλοποιηθούν τα κριτήρια από πλευράς Κομισιόν και η διαδικασία αίτησης ε, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία κρίση και δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Καλό θα ήταν η έκθεση να περάσει λοιπόν με αυτή τη μορφή με τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Κνούτε. Ποιον έχουμε μετά. Χούπναρ. Δεν ζήτησα το λόγο. Αλλά αφού μου δίνετε το λόγο θα ήθελα να πω τα εξής. Η ομάδα του ΕΛΚ σε συνεργασία και με τους φιλελεύθερους και συναδέλφους από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Ε, πάντων, θα μιλήσω εγώ για το ΕΛΚ. Δεν βρήκαμε τις συμβαστικές λύσεις ε, που προτείνει ο κύριος Φέντελ να πλησιάζουν ε, τη συνένεση που θα θέλαμε δεν θεωρούμε δηλαδή πως ε, μας βοηθούν τόσο, οπότε θα επιμείνουμε στην ε, τελική ψηφοφορία σε ε, τα ζητήματα εκείνα τα οποία είχαμε αναφέρει αρχικά στις τροπολογίες μας, γιατί φοβόμαστε πως οι τελικές συμβαστικές τροπολογίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες στήριξης των διαρθρωτικών αλλαγών και του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προς ε, περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Και το ξέρω και εγώ και ο κύριος Χέντελ, απλά θα ήθελα να επαναλάβω πως ε, έχουμε κάποιες έτσι, διαφορετικές ιδέες εμείς, ε, οι οποίες κατά την απόψή μας δεν περιέχονται στις συμβαστικές λύσεις όπως προτάθηκε από τον κύριο Χέντελ. Ευχαριστώ. Θα θέλατε κι εσείς να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ προσωπώ την κυρία Πόδηματά εδώ πέρα που συνεισέφερε σε αυτή την έκθεση. Κυρία Χίμπνερ, εκτιμώ το έργο σας εδώ και καιρό. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στις διαπραγματεύσεις. Ε, απλά εγώ ενημερώθηκα για το ότι εκπροσωπείται τρεις ομάδες. Δεν ξέρω γιατί έτσι και γιατί δεν μπορέσαμε να οδηγηθούμε σε μια συνένεση. Ίσως αργότερα για να μην επαναλαμβάνεται αυτή η κατάσταση. Προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τον εισηγητή γιατί συμφωνούμε με την άποψη. Η κυρία Αποδηματά θεωρεί πολύ σημαντική την έκθεση και συνεισέφερε για να ξεκαθαρίσει πως ε, δεν μιλάμε για βιομηχανική πολιτική ή για πολιτική για συγκεκριμένες εταιρείες όταν χρησιμοποιείται αυτό το ταμείο, αλλά το ταμείο αυτό πρέπει να έχει διαρθρωτικές σε επιπτώσεις, ε, να δημιουργήσει δηλαδή διαρκείς ε, συνθήκες ε, αγοράς εργασίας σε μια περιοχή και έτσι άρα να συμπληρώνει και τους στόχους στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 για να έχει ένα υφόρο διαρκές αποτέλεσμα. Όχι μόνο δηλαδή πυροσβεστικό αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω είναι το κοινό νήμα των συνεισφορών της κυρίας ε, Πόδηματά. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη αυτή η έκθεση. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε κάτι. Γιατί πρόκειται για κάτι σημαντικό για την Επιτροπή μας. Περβάνς. Euh, Ευχαριστώ. Πρόκειται για μία έκθεση που κάνουμε με την Επιτροπή Προπολογισμών, σημαντική γιατί δίνει κάποια, στέλνει κάποια μηνύματα στην Ευρωπαϊκή ναι. Επιτροπή ναι, ναι, όσον αφορά την ουσία. Αν δούμε την αξιολόγηση για το ταμείο αυτό, Υπάρχει ένα σημείο που βέβαια εγώ δεν έχω εδώ μπροστά τα διάφορα, τις διάφορες προτάσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα πολύ σημαντικό σημείο και το λέω γιατί έχει να κάνει και με τροπολογίες της κυρίας Σούμπνερ και είναι το θέμα της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου στις επιχειρήσεις όσοι απολύονται θα πρέπει να μπορούν να υποφελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Στην Ιρλανδία βλέπουμε σε τι βαθμό, άπαξ και δεν υπάρχουν κοινωνικοί εταίροι που να συμμετέχουν στη διαδικασία, σε τι βαθμό λοιπόν ε, χάνουμε. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή καλά. Ε, δεν μπορούμε να υποφεληθούμε αρκετά από το Ευρωπαϊκό Αυτό Ταμείο. Ενώ αντίθετα στην Αυστρία, στη Γερμανία, όπου συμμετέχουν από την αρχή μέχρι το τέλο τη διαδικασία οι κοινωνικοί εταίροι, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Στην Ιρλανδία δεν πάνε τα πράγματα καλά, ακριβώ γιατί δεν υπάρχει συνδικαλιστική δομή τέτοια που να μπορεί να υπάρξει διάλογος των συνδικάτων με τις αρχές. Οπότε εδώ νομίζω ότι η αρχική διατύπωση του εισηγητή στην παράγραφο 5 μάλιστα πρέπει να διατηρηθεί. Και ελπίζω τελικά να συμπεριληφθεί στην τελική γνωμοδότηση που θα ψηφίσει η δικιά μας Επιτροπή. Ευχαριστώ. Is there Άλλος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ για αυτή την έκθεση έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες προκειμένου να αλλάξει λίγο το ύφος της έκθεσης που έχει δύο στόχους η προσπαθιά μου. Ε, ο ένας είναι ότι το ύφος αυτό νομίζω ότι δεν, ήταν, ε, δεν διέπεται από ακρίβεια νομικά και από την άλλη μεριά υπήρχαν και κάποια αντιφατικά στοιχεία κατά τη γνώμη μου γιατί από τη μια ζητούσε ε, πιο συχνή κινητοποίηση του Ταμείου αλλά από την άλλη μεριά με κριτήρια τα οποία οποία δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κινητοποίηση του Ταμείου. Γι' αυτό εγώ θέλω να απλοποιηθεί. Και αυτό ισχύει για όλα τα ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πιστεύω ότι στην επόμενη έκθεση που θα κάνει, την ετήσια ή στην αξιολόγηση την ενδιάμεση που γίνεται, να προτείνει ένα προβληματισμό για τα κριτήρια. Με στόχο πρώτον το ταμείο να αποτελεί πραγματικά πρόσθετη αξία, πέρα δηλαδή από τα διαφορετικά ταμεία, να είναι κάτι παραπάνω, και από την άλλη μεριά να αποτελεί και ένα χρήσιμο μέσο που να μας βοηθάει να δίνουμε απαντήσεις, να ανταποκρινόμαστε στις κρίσεις που μας πλήττουν. Ευχαριστούμε. λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Κλούτε, θέλετε να πείτε κάτι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα στο τέλος για να κλείσει η συζήτηση. Όχι, νομίζω ότι υπόθηκαν ότι ε, πρέπει να υποθούν. Παρακαλώ να υπερψηφίσετε το συμβιβασμό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Και για τίποτα άλλο, περάσουμε στην ψηφοφορία, αν χάνουμε χρόνο.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 Right, everybody, have we, have we got... Χαίρετε, καρτούλες έχουμε. Έχετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε. Um... Να κάνουμε μια δοκιμαστική παρακαλώ ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα ηλεκτρονική. Μια ψηφίσατε όλοι. Wait, wait, where's he gone? He's there. He's there. Where? There. Standing over there. Oh. Right, we're closing the voting. Πέρας. Well, at the moment we've got more cards plugged in than people voting, but uh, I don't think it looks like anybody's over quota at the moment. Λοιπόν, εντάξει, δεν νομίζω να υπερσέβει κανεί. Θα μετράμε, θα βλέπουμε και θα ελέγχουμε και θα σα πούμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεση του κυρίου Κάρα για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Και η πρώτη ψηφοφορία για τροπολογία 2, παρακαλώ ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 23. Παρακαλώ ψήφι υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα. 23 παρακαλώ τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. A Πέρας. Α, καταπίπτει ισοψηφία. Ορίστε κυρία Λούλινγκ. Ε, έρχεται η κάρτα μου, είναι καθοδόν, τώρα φτάνει. Uh, Καταφέραμε να καταψηφιστεί χωρίς εσάς. It falls anyway. Έτσι και με ισοψηφία. 19 κατά λέει η κυρία Λούλη. Δεν πειράζει, 18 φτάνουν. Και προχωρούμε. Στην 24. Ψήφι περ Κατά αποχές ε, γκρίνεται. 25. περ Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παρθμό 4 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να το ελέγξω. 28 παρακαλώ, αρχίζει ψηφοφορία τώρα. Πέρας, εγκρίθηκε. Η τροπολογία υπέρθυμα 5, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30, προφορική τροπολογία εδώ του εισηγητού για να αλλάξουν κάποιες λέξεις και ένα και να γίνει συμπεριλαμβανομένων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 έχει αποσυρθεί. Η 8 ψηφίπε κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Τώρα, στην τροπολογία 9 έχουμε προφορική τροπολογία με μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής που λέει να εξαιρεθούν οι λέξεις, να κατανομαστούν ε, οι υπεύθυνοι, τα υπεύθυνα μέρη. Δηλαδή η προφορική τροπολογία θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει πώς η συλλογή και αξιολόγηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων από τα κράτη-μέλη διεξήχθη στο παρελθόν και να εξαγάγει τα ε, σχετικά συμπεράσματα τα οποία θα αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η νέα προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. είναι η προφορική τροπολογία χωρίς τις τέσσερις λέξεις στα αγγλικά name the responsible parties. Υπέρ, κατά, αβουχές Μα έχετε βερδέψει. Με την προφορική τροπολογία ελέγχουμε λοιπόν, όπως σας είπα, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα ανοίξετε την ψηφοφορία σας παρακαλώ. Εξαφανίστηκε ο Ντόλφο.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 Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται, ωραία. Συνεχίζουμε. Ε, πάμε στην αιτιολογική σκέψη 3. Ψήφι υπέρ της 10. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά άποχες. Θέλετε να ελέγξουμε τη 14 παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. 15 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 16 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 17 είπε. Α, συγγνώμη, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτό το δεύτερο. 18 σύφ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά Καλύτερα να το εγκρίνουμε. Δεν είναι σαφές. Ψήφισατε όλοι. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά το κείμενο, παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. 38-1 με μία από εκεί. Συγχαρητήρια κύριε Κάρας. Και τώρα... Εκλά. Μπορείτε μέχρι και να χειροκροτήσετε. Um, I thought at least I got one with the rapporteur on this. Okay. Okay. Um, this is now the draft resolution Λοιπόν, και πάλι σχέδιο ψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το μηχανισμό. Όχι, συγγνώμη, είναι το Ευρωπαϊκό Μέσο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτική Σταθεροποίηση και Μελλοντικέ Δράσει. Ψήφι Α, ο μπλοκ μέχρι πού όλα αυτά μαζί. Ε, όλες τις αιτιολογικές σκέψεις μαζί δηλαδή. Συγγνώμη, Περβάνς, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ναι, μπορούμε να ψηφίσουμε ένα μπλοκ μέχρι την παράγραφο 3, όλες μαζί. Μάλιστα. Πιο αργά. Όλες οι αιτιολογικές σκέψεις μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί όλο αυτό που αρχίζει having regard. Those in favor, against, abstentions. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τώρα έχουμε την παράγραφο Α9, ε, S&D, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται έλεγχος για την παράγραφο α νέα. Oh, yeah. Thank you. Okay. And that's carried 21-19. 21-19, εγκρίνεται. Η παράγραφος αλφα-αλφα, νέα, ψήφι πέ. Κατά. Απόχες. απορρίφτεται. Παράγραφο α. Ψήφι υπερ... Τι θέλετε έλεγχο για την α. Ψήφισατε όλοι. Απορρίπτεται λοιπόν η ΑΑ. 22 κατά 19 υπέρ. Ερχόμαστε λοιπόν στην παράγραφο α. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα Παράγραφος Β. Με την τροπολογία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είπε Κατά. Τα έχω χάσει εντελώς. No, it Ξαναγυρίστε σας παρακαλώ στην παράγραφο Β. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος C. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δι. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση των πρασίνων στην παράγραφο 1. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην παράγραφο 2 με τροπολογία του ΕΛΚ ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην παράγραφο 2α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και παράγραφος 3 ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν η εκδοχή του ΕΛΚ, αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία των σοσιαλιστών και δημοκρατών υπέρ, γιατί είναι προσθήκη. Κατά αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε, σας παρακαλώ πολύ. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω, μην ανησυχείτε. 3α ε, νέο ψηφίδε κατά αποχές εγκρίνεται ε, παράγραφος 4 με προφορική τροπολογία σοσιαλιστών και δημοκρατών για να αλλάξει η ανταγωνιστικότητα είναι βασικά μια γραμματική διαφορά τροποποίηση γλωσσική. Μάλιστα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 τώρα. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Με τροπολογία και δημοκρατών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8. Το ΕΛΚ την έχει αποσύρει. 8 του φιλελευθέρων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9β σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ο παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές. Παράγραφος 9. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. S&D. Πρώτα. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ηλεκτρονικά. Νομίζω θα είναι πιο εύκολο για μας. Ψήφισατε όλοι. Θα ψηφίσετε όλοι. Απορρίπτεται. Και ερχόμαστε στην αρχική παράγραφο 9. Ψήφι πέ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Το βρασίνο Υπέ. Κατά αποχές μπορούμε να το αλλάξουμε, παρακαλώ τα 11 Μου ψηφίσατε όλοι, απορρίπτεται. Έντεκα εισεντή υπέρ, κατά, αποχές, επίσης απορρίπτεται. Παράγραφος 11, η εκδοχή του ΕΛΚ είπε, Κατά. Αποχές. Και αυτό νομίζω έχει απορριφθεί. Αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα. Η 11 του ΕΛΚ. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Μάλιστα. Και προχωρούμε στην παραγραφό 11α νέα των πρασινων ψήφιπε κατά υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. 11β νέα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές. Μπορούμε σας παρακαλώ να το ελέγξουμε αυτό. Το πρώτο τμήμα της 11β. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. Και το δεύτερο καταπίπτει. Ωραία. Ε, προχωρούμε στη 12 του σοσιαλιστών. Ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12α. 9 με προφορική τροπολογία. Αν ψηφίσουμε αυτή, καταπίπτει η αρχική. 12α νέα προφορική τροπολογία. Που μιλάει για τα ευρωομόλογα. Ότι είναι συμβατή με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη, ενώ το αρχικό κείμενο λέει κάτι διαφορετικό. Υπέ, Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο ελέγξουμε παρακαλώ. Yes, that, was carried. Εγκρίθηκε. Ωραία. 13 S&D Ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η αρχική παράγραφος 13 επέν Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 14. Παρακαλώ. Α, όχι 14, δεν γίνεται. Καλά, θα τους το πούμε. Ε, το κείμενο όπως τροποποιήθηκε παρακαλώ κατευθείαν ηλεκτρονικός. Somebody being slow, one more to come. Okay, no, everybody voted who's going. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Now move on. Τώρα συνεχίζουμε. Και περνάμε στην χρηματοδότηση του Τόμα Σέντελ για τη χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Είσαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία Α. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Συνεπώς, η 1 έχει αποσυρθεί, η 2 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Οι άλλοι για το 1-1 καταπίπτουν και πάμε στην τροπολογία 5. Υπέρ παρακαλώ. Για την παράγραφο 5, έτσι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στις τροπολογίες Τροπολογία 6 και 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Οι υπόλοιπε μέχρι την 11 καταπίπτουν. 11 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Γ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες τώρα 12, 13 και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία δέλτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίνεται, γιατί απέχει το έλκα, αλλά να ελέγξουμε αν θέλετε. Είμαστε στην τροπολογία 17. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ζαμπόλ. Εκτός μικροφώνου, δεν ακούγεται. Η 16 απορρίφθηκε, την ψηφίσαμε. 17 τώρα. 17. Ελέγχουμε για την τροπολογία 17. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 και 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ για τις 19 και 20. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της προφορίας, εγκρίνεται. 21 ε, πίπτη, Συμβαστική ε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε τώρα στην τροπολογία 26. Υπέρ παρακαλώ της 26. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ για την 26. Πολύ παρόμοιο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο, παρακαλώ ηλεκτρονικά όμως. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή λοιπόν. Δεν έχουμε άλλες ψηφοφορίες. Οπότε συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο θέμα. Αριθμός 9. CRD 4. Βασιλεία 2. Is one of you taking the chair for this or not? I wasn't asked to. I've got CRD Yeah. Um, um,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 Λυπάμαι, συγγνώμη συνάδελφοι, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ πέρα και υπάρχει και άλλος ένας ε, τριμερής ε, διάλογος, ε, εδώ στον οποίο πρέπει να πάει η πρόεδρος. Τέλος πάντων βρήκαμε έναν αντιπρόεδρο και πιέζει και ο χρόνος. Okay. <laughs> Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στην συζήτηση της έκθεσης του κυρίου Κάρας. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ πέρα να συζητήσουμε την έκθεση για την τέταρτη οδηγία σχετικά με την κεφαλιακή επάρκεια ή γνωστή και ως Βασιλεία 3. Οπότε πριν περάσω στις ε, τροπολογίες να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. ο εισηγητής θεωρώ την απόφαση των G20 για την Βασιλεία 3 λανθασμένη αντιπαραγωγική και επί της ουσίας και πολιτικά αποτελεί υπεκφυγή από τις ευθύνες μας. Πριν συμφωνήσουμε στη Βασιλεία, στη Συμφωνία, οι G20 διαπίστωσαν και όρισαν πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και δεύτερον πως μπορεί να υπάρξει μεμονωμένη εφαρμογή και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κοινή η εφαρμογή. Δηλαδή αυτό δεν είναι απάντηση στην κρίση. Γιατί αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ίση όροι ανταγωνισμού και να μην υπάρχουν ανισότητες και να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο για να μην έχουμε περαιτέρω στρεβλώσεις. Το να δηλώνουμε πως θα γίνει αλλά δεν ξέρουμε πότε και πώς και δεν μας νοιάζει πώς θα εφαρμοστεί και ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, ε, δεν είναι πολιτική ευθύνη και δεν ανταποκρίνεται και στην ουσία της ε, κεφαλιακής επάρκειας ως απάντηση στην Κρήτη. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο να ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το χρονοδιάγραμμά μας. Βεβαίως για εμάς σημασία έχει ουσία και όχι το χρονοδιάγραμμα και θέμε μια ουσία με την οποία θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και αφού συμφωνήσουμε σε αυτό θα δούμε το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής. Και να υπενθυμίσω πως έχουμε δύο αποφασιστικά σημεία εδώ πέρα στην έκθεση αυτή. Το πρώτον πως εμείς θεωρούμε πως η Βασιλεία και η Επιτροπή πριν ληφθεί απόφαση και γραφτεί οδηγία θα πρέπει να κάνει μια μελέτη για τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία γιατί βεβαίως αυτό εδώ πέρα δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μέσο οι τράπεζες για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Δεύτερον αυτό το οποίο απαιτούμε να δούμε το σορευτικό αποτέλεσμα των υπαρχόντων μέτρων στις χρηματαγορές όσον αφορά την επίδρασή τους και να γίνει μια σούμα τελικά. Γιατί έχουμε κεφαλαιακή επάρκεια 3, κεφαλαιακή επάρκεια 4, μιλάμε για φόρο συναλλαγών, μιλάμε για τραπεζικές εισφορές και αυτά τα οποία έχουμε και σε σχέση με την ασφάλιση, την, εγγύηση των καταθέσεων. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, να δούμε τι γίνεται και με την πραγματική οικονομία και όπως σας είπα με τα σωρευτικά αποτελέσματα όλων αυτών. Και όλα αυτά είναι κομμάτι της έκθεσής μας. Κατά την άποψή μου, μέσω της απόφασης των G20 δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε κανόνες που είναι ουσιαστικά σημαντικοί κατά την άποψή μας και θα πρέπει να τονίσει τη διαφορά μεταξύ τραπεζικών δομών ΙΠΑ και Ευρώπης. Και ακριβώς λόγω των εξελίξεων στους G20 αποδίδω εγώ ιδιαίτερη πολιτική σημασία σε αυτό. Πρέπει να αντιληφθούμε την ευθύνη μας. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες 258 τον αριθμό, κάτι το οποίο δείχνει πως αξίζει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα και δεν πρόκειται μάλιστα για νομοθετική έκθεση αλλά για ένα πολιτικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οκ, okay, ε, βεβαίως αυτές οι 258 απολογίες ε, καταδεικνύουν πόσα ερωτήματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν στην Κομισιόν και στην Βασιλεία για να οδηγηθούμε σε κάποιες εξελίξεις. Το μεγαλύτερο κομμάτι των ε, τροπολογιών πηγαίνουν προς την κατεύθυνση του σχεδίου έκθεσης και όπως αντιλαμβάνεστε λόγω του ορίου του αριθμού των λέξεων δεν μπόρεσα να μπω σε λεπτομέρειες αλλιώς εγώ πολύ ευχαρίστος να έχουμε τροπολογίες και να εμπαθύνω αλλά διαπιστώνω πως ε, πρέπει να κάνουμε μια διάρθρωση. Τώρα θα μιλήσουμε για την πολιτική πτυχή και δεν έχουμε μπει ακόμα σε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για την οδηγία. Γι' αυτό εγώ θέλω να ενισχυθεί η πολιτική πτυχή της έκθεσης ακριβώς ως απάντηση στους G20 και όχι οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις. Εκεί θα βοηθήσουν πάρα πολύ αυτές οι συμπληρώσεις. Στόχος πρέπει να είναι ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους και ίδια εφαρμογή. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος εφαρμόζει τελευταίος να ωφελείται κιόλας. Δυστυχώς γι' αυτό πρέπει να, να δράσουν οι G20. Αυτό το οποίο αποφάσισαν εκεί πέρα είναι για μένα ανεξήγητο. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων, νομικών μορφών και δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέφερε ήδη να γίνει θέμα η κεφαλαιαρκή επάρκεια 4, αν και εγώ δεν θεωρώ πως δεν είναι έτοιμη προς απόφαση στην Επιτροπή της Βασιλείας, οπότε δεν είναι έτοιμη για απόφαση στην Κομισιόν. Και αυτή θα έπρεπε να προτιμήσουμε αντί για απόφαση της Βασιλείας. Και τα δύο αυτά δεν τα θεωρώ δεδομένα. Δεν θεωρώ πως υπάρχουν προϋποθέσεις για απόφαση στην Επιτροπή της ε, Βασιλείας ε, καθώς και για το τι αναμένουμε μετά ως ε, πρώτος οδηγίας μετά την απόφαση των G20. Όλοι αναφέρονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές τις τροπολογίες τις στηρίζω. Πράγματι πρέπει να γίνει μια μελέτη επιπτώσεων. Επίσης, εγώ είμαι ανοιχτός για το ότι η Κομισιόν θα πρέπει να παίξει σημαντικότερο ρόλο και πρέπει τώρα να συντονιστεί καλύτερα με το Κοινοβούλιο για να συντονιστούν τα κράτη στην Επιτροπή της Βασιλείας. Νομίζω πως υπάρχει συμφωνία για το ότι τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό κομμάτι και τα νομικά δεν μπορούν να αποτελέσουν το αποφασιστικό κριτήριο, αλλά η ποιότητα του, ε, της κεφαλαίκης επάρκειας. Έχουμε τρεις νομικές μορφές, επενδυτικές τράπεζες, ανώνυμες εταιρείες και λιανικές και τράπεζες τραπεζικής λιανικής Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα μπορούν να διατηρηθούν βιώσιμες, να απορροφήσουν τα κέρδη, τα, τις ζημίες με συγχωρείτε, και το ζήτημα βεβαίως του δανεισμού. και βεβαίως πώς ε, ανταποκρίνονται σε διάφορα, διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Οπότε η σταθερότητα του συστήματος είναι ο κύριος ε, στόχος. Πρέπει να δούμε επίσης το τι γίνεται όσον αφορά στη διαφορετική αντιμετώπιση στοιχείων του υπολογισμού και των παραγόγων. Το ίδιο ισχύει και για τη διαφορά μεταξύ φορολογικών ε, ισολογισμών και άρα υπάρχει και ο κίνδυνος ε, συγκέντρωσης ο οποίος θα πρέπει να εμποδιστεί και ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους. Επίσης όσον αφορά τη μόχλευση υπάρχει ο κίνδυνος να πληγεί χειρότερα η Ευρώπη από ότι άλλοι συμμετέχονται στην ε, αγορά καθώς είναι χαμηλότερος το ποσοστό μόχλευσης. Όλες Αυτές οι διαφορές δεν γίνονται με μια προσέγγιση one size fits all, να λάβουμε δηλαδή μέτρα τα οποία θα ισχύουν για όλους. Ε, θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ποιο θα είναι το στόπο στο και μετά να μιλήσουμε για πυλώνα 1 ή πυλώνα 2. Νομίζω πως υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν συμβασμοί με αυτούς που κατέθεσαν τροπολογίες. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τους σκιώδεις ηγητές να κάνουμε μία συζήτηση, να υποβάλουν συμβαστικές προτάσεις και ελπίζω μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου να εκμεταλλευτούμε το χρόνο για να συνεννοηθούμε είτε τηλεφωνικά είτε με email για να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία στις 6 Σεπτεμβρίου και σας ευχαριστώ για την επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστούμε κύριε Κάρας. Θα ήθελα εγώ τώρα να, να ζητήσω από τους συναδέλφους να παραμείνουν στα χρονικά όρια, στο όριο των τριών λεπτών. Γιατί έχουμε άλλα τρία, τρεις εκθέσεις. Θα δώσω τον λόγο λοιπόν στους και κύριος Μπούλμαν πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μπορώ να τα καταφέρω σε τρία λεπτά, αλλά ε, ξεκινήστε το ρολόι τώρα που έχει τη δυνατότητα να με ακούει και ο εισηγητής συμφωνώ με την εκτίμηση του συναδελφού Κάρας για το πώς χειριστήκαμε καταστροφικά αυτό το θέμα στο Τορόντο. Δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο το να μην έχουμε λογικές απαντήσεις, το να αναβάλουμε συνεχώς. Δεν ενισχύεται έτσι η οικονομία, ούτε η εμπιστοσύνη του λαού στην πολιτική και στο αν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Και Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί έχουν έτσι τα πράγματα. Ξεκίνησε νομίζω και η συζήτηση με τον κύριο Σέμετα με αυτό. Νομίζω πως οι Ευρωπαίοι δεν ε, στέλνουμε ξεκάθαρα μηνύματα για το τι θέλουμε και από τους άλλους και από μας. Και Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν, συμφωνούμε και με αυτό, να αναμειχθεί ενεργότερα στη Βασιλεία και να μας λέει και το τι κάνει εκεί πέρα. Και να συζητάει και πιο διάφανα με τα κράτη-μέλη. Τα οποία και αυτά πρέπει να προχωρήσουν σε κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Αλλά εάν δεν γίνει κάτι τέτοια, μην παραπονιόμαστε μετά για το ότι δεν έχονται και άλλοι μαζί μας. Και έχει δίκιο ο κύριος Κάρας όταν λέει πως πρέπει να προσέξουμε με τους νέους κανόνες να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις στις οποίες κάποιοι θα εκμεταλλεύονται τις διαφορές ε, της νομοθεσίας ε, και ε, θα έχουμε έτσι στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Ένα πράγμα όμως μας χωρίζει και δεν ξέρω, θέλω να δω εάν μπορούμε να συμβαστούμε τις ερχόμενες εβδομάδες. Όταν εμφανιστεί ένα πρόβλημα στο μέλλον, δεν οφείλεται αυτό μόνο στις ε, τράπεζες. Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία των κανόνων, οπότε πρέπει να δούμε και ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Και εγώ δεν θεωρώ, και αυτή είναι η τελευταία και σημαντικότερη σκέψη μου, δεν θεωρώ πως λόγω των στρεβλώσεων αυτών του ανταγωνισμού που φοβόμαστε να μην κάνουμε καθόλου μεταρρυθμίσεις όταν πρόκειται για να γράψουμε τους δικούς μας κανόνες κεφαλαίκης απέτηση. Το αντίθετο, το αντίθετο. Η κεφαλαϊκή επάρκεια 3 δεν θα λύσει τα πάντα, θα παραμείνουν πολλά πράγματα απ' έξω, αναφέρω τα στοιχεία εκτός ολογισμού, την αντικυκλική εγγύηση που δίνουμε. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτό στο πακέτο, αλλά χρειαζόμαστε το να προχωρήσει επιγόντως η μεταρρύθμιση του πακέτου της κεφαλαιακής επάρκειας και να μην τα παρατήσουμε γιατί κολλάμε στο διεθνές επίπεδο. Είτε όλοι μαζί, είτε ε, κανένας δεν νομίζω ότι είναι ως κανένας. Εμείς θέμε να συνεχίσουν να μεταρρυθμίζονται οι τράπεζες και βέβαια να λειτουργούν αυτό εννοείται. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Φόρντ, επίσης και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καρά και όλους τους συναδέρφους που υπέβαλαν ε, τόσες τροπολογίες. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας ότι το σημαντικό είναι το χρονοδιάγραμμα, το πότε γίνονται όλα αυτά, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να βρεθούν στη σωστή στιγμή του κύκλου και να αναγνωριστούν τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Αλλά να υπάρξει επίσης και διεθνή συμφωνία. Πολλά από αυτά τα είπαν το Σαββατοκύριακο οι G20 και αντικατοπτρίζονται και στα σχόλια των συναδέρφων μέσω των τροπολογιών τους. Πράγμα που δείχνει ότι είναι το θέμα πιο πολύπλοκο από ό,τι νομίζαμε. Όπως το λένε και οι 20. Τα σχόλια του κύριου Πόλμαν πιστεύω ότι είναι πολύ καλά. Για το θέμα των δοκιμών. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την άποψη του κυρίου Καρά εδώ, ότι οι δοκιμές αυτές πρέπει να υπάρχουν όπως τις έχουμε προβλέψει με πολύ διαφάνεια για τα παράγωγα. Και εδώ υπάρχουν καλά στοιχεία για clearing, για τυποποίησεις, πράγματα που είπαν και οι G20 και πρέπει να φροντίσουμε ότι μερικές φορές ορισμένοι χρειάζονται διαφορετικά παράγωγα από τράπεζες που έχουν το μεγαλύτερο κεφάλαιο και δεν θα πρέπει να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο δυσμενής μεταχείριση όταν φτάνουμε στην πρόσβαση στην αγορά και στα κεφάλαια. Πάντως εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μία λύση για όλες τις περιπτώσεις, για τους ρυθμιστές, τους επενδυτές, ε, για εκείνους που συλλέγουν τους φόρους. Μπορούμε να κάνουμε κάποια διαφοροποίηση. Επίσης, πολλά σχόλια ακούσαμε για τον δίκτυ μόχλευσης. Είναι προφανές ότι όντως υπάρχει υψηλή μόχλευση. Ας φροντίσουμε λοιπόν να μην μιλήσουμε για τον έλεγχο του τελικού να μιλήσουμε καλύτερα για την συμμετοχή. Να δούμε δηλαδή τι λύσεις υπάρχουν, ακόμα και αν είναι δύσκολες. Για τη ρευστότητα, ναι, πρέπει να μειώσουμε τους κινδύνους συγκέντρωσης. Αλλά πρέπει επίσης να έχουμε και κεφάλαια ρευστού. Και κατά τα για τη, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία πιστεύω ότι Οπότε η τετλοποίηση, όπως λένε και οι Financial ties, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να κλείσουμε από τώρα, πρέπει να δούμε όλες τις λύσεις που υπάρχουν για το νέο κεφάλαιο και για την ποιότητα του κεφαλαίου. Κάποιοι λένε ότι οι αλλαγές όσον αφορά τους τύπους κεφαλαίων πρέπει να πάνε πολύ μακριά. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν σφάλμα κάτι τέτοιο. πρέπει να φροντίσουμε οι απώλειες να λαμβάνονται υπόψη, αλλά αυτό πριν φτάσουμε να έχουμε το χρήση της τράπεζας ή μια τράπεζα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Ο κύριος Κλούτε τώρα. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Ήδη υπόθηκαν πολλά και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω και εγώ άλλωστε. Έχουμε υποβάλει μερικές τροπολογίες εξ ονόματος της ομάδας μου με στόχο κυρίως να οξύνουμε κάπως τη διατύπωση, ε, να προχωρήσουμε τα πράγματα και στα πλαίσια των συμβαστικών τροπολογιών θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Λάμπερτς είναι σκιώδης ηγητής, αλλά δεν το γράφει εδώ ο κατάλογος των αγορητών. Παρακαλώ. Καλώς. Λοιπόν, Καταρχάς, για το πολιτικό περιεχόμενο συμφωνώ πολλά με τα όσα υπόθεσα. Είναι ολέθριο παράδειγμα του G20 για το προς αποφυγή όλες. Και θα πρέπει το συντομότερο να φέρουμε δική μας νομοδότηση. Και έχει σημασία να συμφωνεί η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Η σημερινή εμπειρία της εποπτείας σε πολλά θέματα την Ατζέντα 2020 δείχνει ότι για να ακουστεί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει μία φωνή. Και έτσι θα αποδείξουμε και στο Συμβούλιο ότι υπάρχει δυνατότητα όντω να έχει μία φωνή το Κοινοβούλιο ε, με συντριπτική πλειοψηφία διαφόρων πολιτικών ομάδων και διαφόρων χωρών που εκπροσωπούνται εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό από μόνο του ε, να το πράξουμε αυτό και η ταχύτητα, και συμφωνώ με τον κύριο Κάρα, είναι επίση σημαντική. Μερικά σημεία μόνο. Ακούμε τώρα τις τράπεζες να λέγουν ότι προσοχή να δούμε με ποιο τρόπο θα εισαχθούν τα διάφορα μέτρα που προγραμματίζουμε σταδιακά. Δεν θα τα ακούμε, εντάξει, αυτό το λένε οι τράπεζε, αλλά βάλουμε εμεί όρου και προϋποθέσεις. Εάν εισάγουμε προοδευτικά με προγραμματισμένο τρόπο κάποια πράγματα, θα πρέπει να δεχθούν συμπληρωματικούς ε, περιορισμούς ε, οι τράπεζες, για παράδειγμα περιορισμό των αμοιβών των στελεχών τους, των διευθυντικών και ε, τα μερίσματα και τα μπόνου που δίνουν στου μετόχους. Αν μας ζητούν εμά να είμαστε επίκης και σιγά σιγά να βάλουμε μέτρα, τότε και θα πρέπει να βάλουν και αυτοί νερό στο κρασί τους. Δεν μπορούν με τρόπο παράλογο να ε, αμείβουν και στελέχη και μετόχους. Και σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, το βασικό είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, κύριε Κάρας, να ξανάρθει στο πραγματικό του ρόλο, να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Αλλά να γίνει αυτό, θέλω να το δω στην πράξη. Μα ζητούν βαθμοί να εισάγουμε νέα μέτρα, αλλά θα πρέπει και εκείνοι να αποδείξουν ότι χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Και αυτό δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε επαρκή βαθμό. Δεν θέλω να επανέλθω στην ουσία πολλών τροπολογιών που υποβάλαμε. Και ένα τελευταίο. βεβαίω θέλουμε ίσους κανόνε παιχνιδιού, αλλά αυτό είναι κάτι το ιδεώδες. Εντάξει, στη πράξη δεν υπάρχει, είναι οτοπία. Γιατί ο πλανήτης ε, έχει τρομερές διαφορές. Και θα έπρεπε να το είχαμε πει και στο Τορόντο ότι θέλουμε παγκόσμια μέτρα, αλλά και να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία και σε αυτή την περίπτωση και για το φόρο των συναλλαγών, ότι αν δεν γίνει αυτό, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, θα συνεχίσει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό να είναι το σαφές μήνυμα. Δεν υποθηκεύουμε το μέλλον μας ε, όμοιρο στα χέρια μιας υποτιθέμενης ε, παγκόσμιας προσπάθειας που θα έρθει μετά από δεκαετίες. Ο κύριος Λούλινγκ λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω πόσο συμφωνώ με τον εισηγητή μας και την εισαγωγή του διότι αυτά που συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφή στον 20ο Τορόντο το Σαββατοκύριακο, ή μάλλον τα όσα δεν συνέβησαν, είναι ενδεικτικά. Και τονίζουν ακόμα περισσότερο αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι τους επόμενους μήνες σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των χρηματαγορών. Παρόλο που ορισμένοι κάνουν πιο προσπάθειες, οι βασικές οικονομικές δυνάμεις βγαίνουν από την κρίση ασύντακτα, ατα, ατάκτος. Είναι πολύ λίγος ο συντονισμός. Ο ε, κάθε μεγάλος οικονομικός παράγων και κάθε μεγάλη χώρα ε, δρά σύμφωνα με την ίδια της κατάσταση, τις πεπιθήσεις, τις παραδόσεις κτλ. Οπότε εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα όσα πράττουμε ως Ευρωπαίοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό άλλωστε να ε, βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσει σύνεσης που μας υπαγόρευσε η κρίση ε, και τους περιορισμούς, ε, τους υπερβολικούς, τους κορσέδες δηλαδή που θα οδηγήσουν σε ασφυξία ε, τον κλάδο και θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας στον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Όχι όλα, αν δεν είναι όλοι στην ίδια μοίρα, ή, αν δεν είναι οι ίδιοι οι κανόνες παντού, αυτό μπορεί να είναι ολέθριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, να έχει συγκριτικό, ας πούμε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα η Ευρώπη. Για τις τροπολογίες, συμφωνώ πολύ με τις ανησυχίες του Ότμαρ Κάρας περιορίζομαι να διευκρινίσω λίγο για τη μόχλευση. Έχω βάλει μια ιδέα, προσπάθησα, ε, που να αφορά μόνο τις επικίνδυνες ή ε, κερδοσκοπικές ε, τοποθετήσεις ή συναλλαγές. Ε, θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτή την ιδέα περισσότερο, παρά να βάλουμε ένα ή περισσότερους δείκτες ή ε, κλάσματα ε, ράσιο. Ε, ε, για πραγματικούς κινδύνους ε, και σε ό,τι αφορά τις παραδοσιακές δραστηριότητες που δεν είναι μεγάλο το ρίσκο δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σκόπιμο, αξίζει να το ελέγξουμε, να το μελετήσουμε με την καλύτερη δυνατή προσοχή, όχι μόνο εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα δεύτερο που έχει να κάνει ε, με ε, την τράπεζα των ε, καταθέσεων. Και πάλι φοβάμαι ότι το παρακάνουμε. σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία και κινδυνεύουμε να την ε, παρεμποδίζουμε αυτή. Και οι μελλοντικοί κανόνες ρευστότητας θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις καταθετικές τράπεζες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις, ε, επενδυτικά ταμεία, ε, το cover bonds για τις ε, νυπόθηκες ε, συναλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ο εισηγητής να με ακούσει και να λάβει υπόψη αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, the floor is with uh, Mr. Hockmark. Thank you very much. And, um, Κύριος Χόκμαρκ. That when we discuss είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το νέο σχεδιασμό των διαρθρωτικών ε, πλαισίων. Να έχουμε καθολική προσέγγιση γιατί η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι πολύ περισσότερο από το να εξασφαλίσεις ένα κλάδο της οικονομίας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ε, θα έχουμε ανάπτυξη, σταθερότητα, ενεργητικό και ε, κανονισμούς που όλα αυτά να τα υποστηρίζουν. Καμιά φορά όταν μιλούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη χρηματοοικονομική κρίση, πολύ συχνά ε, επικεντρωνόμαστε στη φερεγγιότητα που γενικά δεν ήταν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Προβλήματα μπορεί να είχαμε στις ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά δεν ήταν το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα ποιο ήταν. Η ρευστότητα και ακόμα περισσότερο η εμπιστοσύνη που υπονομεύθηκε και χάθηκε γιατί δεν υπήρχαν αρκετά σαφείς κανόνες. Είδαμε λοιπόν τι θα πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον, δηλαδή τις ανεπιθύμητες συνέπειες. έγιναν κάποιες αποκαλύψεις, αναγκάστηκαν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες να εκποιήσουν μαζικά και ταχύτητα, με ε, αποτέλεσμα την κατάρρευση. Αυτές οι ανεπιθύμητες λοιπόν συνέπειες ή παρενέργειες είναι σήμερα πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί αν δούμε άλλη προοπτική από αυτή που είπαν οι συνάδελφοι, αν επιστρέψουμε στους G20 και σε Ευρωπαίους ηγέτες και τα όσα είπε το Κοινοβούλιο, τι σημαίνει αυτό, τα επόμενα έτη, την επόμενη δεκαετία δηλαδή, χρειάζεται μείωση ε, των δημοσιονομικών ελλημάτων. Άρα, από αυτή την πλευρά της οικονομίας θα έχουμε συρρήκνωση και δεν μπορούμε ταυτόχρονα να νομοθετούμε με τρόπο που να έχουμε και άλλη ε, συρρήκνωση και ε, στραγγαλισμό ε, των πιστώσεων γιατί και πάλι θα έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες και θα έχουμε άλλου είδους χρηματοοικονομική αστάθεια. Και θέλω να υποστηρίξω και να υπογραμμίσω αυτά που είπε ο, ο εισηγητής για μελέτη επιπτώσεων. Αυτοί οι κανόνες, αυτή η νομοθεσία, τι θα σημάνει για τις ευκαιρίες ε, χρηματοδότησης επενδύσεων και και να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες για την ανταγωνιστικότητα και να είμαστε ηγέτες παγκοσμίω. Και να ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε το σωστό, το, το υπαρκτό, το πραγματικό πρόβλημα και όλοι οι, βανώνες, κανόνες να βασίζονται ε, στην αποτίμηση του κινδύνου. Και είναι λίγο περίπλοκο, περίεργο όταν μιλάμε για τη μόχλευση, για να λύσουμε ένα πρόβλημα που δεν έχουμε στην ουσία, που το έχουμε αντιγράψει από τις Ηνωμένε Πολιτείε και που δεν λειτουργήσε. Δηλαδή, θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που δεν έχουμε με μια λύση που δεν λειτουργεί. Προσοχή λοιπόν, τα ξέρει και ο εισηγητής ε, τι ε, κανόνες θα αποφασίσουμε. Ελλιώς, κινδυνεύουμε να παρεμποδίσουμε την ανάπτυξη και να υπονομεύσουμε τη σταθερότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Περές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ εισηγητά για την πρόταση αυτή, η οποία μας επιτρέπει να καταλήξουμε στην θέση μας πριν είναι πολύ αργά. Πριν βρεθούμε προτελεσμένων γεγονότων και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή για το ότι τα τεχνικά ζητήματα της ρύθμισης είναι πράγματα που θα δούμε και αργότερα. Αυτό που είναι σημαντικό με την έκθεση αυτή τώρα είναι να στείλουμε κάποια πολιτικά μηνύματα. Γι' αυτό και προτείνω στον εισηγητή, και αυτό έκανα και με τις τροπολογίες που έχω υποβάλει, τρία θέματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Το πρώτο καλύπτει μια ανησυχία που ανέφερε και αυτός, που είναι το συνολικό θέμα του το αντικτύπου που θα έχει αυτή η νομοθεσία. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα εδώ που νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν. Όχι ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις τράπεζες, όχι βέβαια, αλλά θέλουμε να επαληθεύσουμε, να δούμε πώς η εξέλιξη αυτή της νομοθεσίας μας στον τομέα των τραπεζών θα ευνοήσει ή όχι τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και συγχρόνως θα έλεγα να προσθέσουμε και άλλα δύο στοιχεία που ελπίζω να σας βρουν σύμφωνους. Το ένα είναι η ιδέα ότι άπαξ και υπάρχουν επενδύσεις, πρέπει να κοιτάμε και με το άρθρο 9 η συνθήκη της Λισαβόνας μας το ζητάει αυτό, να δούμε πώς θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης με τις επενδύσεις αυτές. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να ευνοήσουμε επενδύσεις οι οποίες αντίθετα θα καταστρέφουν θέσεις απασχόλησης αντί να δημιουργούν. Γενικά μιλώντας πάντως, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην απασχόληση. Κάτι άλλο που το είπατε κι εσείς, η Ευρώπη χαίρει μιας διαφοροποιημένης τραπεζικής αρχιτεκτονικής. Ε, στη Βασιλεία, αυτοί που φτιάχνουν τις ρυθμίσεις, δεν έχουν στο μυαλό τους τη διατήρηση αυτής της αρχιτεκτονικής τραπεζικής ποικιλομορφίας που έχουμε στην Ευρώπη. Στην μελέτη λοιπόν καλά θα κάνουμε να κοιτάξουμε τι συνέπειες θα έχει η νομοθεσία σε αυτήν την ποικιλομορφία της τραπεζικής μας αρχιτεκτονικής.